Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Θα είναι σύντομη η συνεδρίασή μας. Ε, ε, le, principe d'une Εδώ και πολλούς μήνες είχε καθοριστεί η ιδέα της ε, συνεδρίασης σε πέμπτες απόγευμα, όταν ακόμα στεκόταν το ταβάνι της Και είχε προβλεφθεί χθε και σήμερα να γίνει μια μήνυ ολομέλεια και κάτα τα Ιωθώτα τις πέμπτες των ε, μήνυ ολομελιών έχουμε, είχαμε μια συνεδρίαση ως Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πέφτον το ταβάνι εξακολουθούμε να έχουμε μια συνεδρίαση. Αλλά έχουμε ακόμα ένα κακό ιονό αυτό το απόγευμα γιατί ο πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων, ο κ. Βέρνερο, ο οποίος επρόκειτο να έρθει για μια ανταλλαγή απόψεων, μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μου τηλεφώνησε στο τέλος του πρωινού για να μου ανακοινώσει ότι είναι κλινήρης, έχει κολλήσει γρήπη και δεν θα μπορέσει να έρθει. Ευτυχώς ο πρόεδρος Σούλτς είναι σε φίνα φόρμα είναι στο Δουβλίνο για να συναντήσει την Ελλαδική Προεδρία, αλλά ο ιός έχει φτάσει πια της γρήπης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις επενδύσεις της. Επομένως, ως συνέπεια του οποίου θα ελαφρύνει ακόμα περισσότερο η ημερήσια διάταξη των εργασιών μας. Είδατε την ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να διαγράψουμε το σημείο υπαριθμών 8, αλλά θα διατηρηθεί το σημείο 7 που είναι η παρουσίαση από την Κομισιόν της διαδικασίας καταμερισμού κινδύνων με τα νέα εργαλεία των λεγόμενων project bonds, των ε, ομολόγων έργων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τελειώσουμε μέχρι τις 4.30. Σχόλια για την της Όχι, έχει εγκριθεί. Τώρα, από την πλευρά του Προέδρου, θέλω να σας κάνω μία ανακοίνωση. Ο συνάδελφός μας Αλεξάνδρ Άλβαρο ήταν θύμα ενός πάρα πολύ σοβαρού ατυχήματος τροχαίου. Είναι στο νοσοκομείο, βρίσκεται σε κόμμα εδώ και πολλές μέρες. Δεν έχω ε, νέα σε σχέση με την κατάστασή του. Ξέρουμε ότι η κατάσταση του είναι πολύ σοβαρή. Και φυσικά θα διαβιβάσω στην οικογένειά του και στους οικείου την έκφραση της συμπαράστασή μας και τις ευχές μας, τις προσευχές μας για την ταχεία ανάρρωσή του, το ταχύτερο δυνατό και την αποκατάσταση της υγείας του. Οι άλλες ανακοινώσεις μπορείτε να τις βρείτε στο Kobo News. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο σημείο τώρα που είναι το διορθωτικό σε σχέση με το ψήφισμα για τις κατευθυντήρες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό το διορθωτικό σημείωμα μας υπευλήθη μετά από μια επιστολή που μας απέστειλαν, απέστειλαν οι πρώτοι δύο πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές σε σχέση με κάποιο σφάλμα το οποίο είχε παρισφρήσει κατά τη διάρκεια της ψήφισης αυτού του ψηφίσματος για τις κατευθυντήρες γραμμές του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2014. Πρέπει λοιπόν να το υποβάλω στην έγκρισή σας, το διορθωτικό αυτό. Θα θεωρήσω ότι εγκρίνεται αυτό το διορθωτικό σημείωμα, εάν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση η οποία θα διατυπωθεί. Ο Γιάνν Μίλντορ ζήτησε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς η φιλελεύθερη ομάδα θέλει να γύρει μια αντίρρηση, γιατί πρόκειται για μια τροπολογία και των φιλελευθέρων σχετικά. Δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία μετά από την ψηφοφορία ο πρόεδρος, ο προεδρεύων τότε στη συνεδρίαση όρισε ότι αυτή η τροπολογία ήταν παραδεκτή και βάσει του κανονισμού δεν μπορεί να ανακληθεί το παραδεκτό μιας τροπολογίας. Ήταν απλώς θέμα να ψηφιστεί υπέρ ή κατά αυτή η τροπολογία. Ωραία. Καταγράφουμε λοιπόν την παρατήρηση του Γιάννη Μιλντορ και της φιλελεύθερης ομάδας. και θέτω σε ψηφοφορία το διορθωτικό. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Ήθελα απλώς να σας πω εν συντομία ότι από την πλευρά της Edith Herzog δεν υπήρχε καμία πρόθεση να τροποποιηθεί η, η ψηφοφορία, αλλά για κάποιους λόγους δεν υπήρχε η πλήρης προσοχή του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας και δεν μπόρεσε επομένω να καταλάβει το ότι είχε γίνει μια αίτηση για έλεγχο ψήφου σε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν το θέμα λοιπόν να αλλάξει η ψηφοφορία. Απλώς είχε εκφωνηθεί με λανθασμένο τρόπο αυτή η ψηφοφορία. Μερικέ φορέ μπορούν οι αντιπρόεδροι να διορθώσουν αυτό το οποίο είπαν. Αυτή τη φορά δεν έγινε και γι' αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό. Καλώς. Αυτό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Υποβάλλω το διορθωτικό σημείο. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τέσσερις, πέντε ψήφι κατά. Αποχές. Η Γκουε, μάλιστα. Οπότε γίνεται δεκτό το διορθωτικό σημείωμα. Αλλά φυσικά αυτό, όπω είπα προηγουμένω, δεν αλλάζει τίποτα από το περιεχόμενο της ψηφοφορία. Παίρναμε τώρα, εάν θέλετε, στο σημείο 6, γιατί ο εισηγητή μα ο κύριο Τόρβαλτ, ε, βιάζεται. Πρόκειται για το συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνα για το σχέδιο ΙΤΕΡ. Έχει το λόγο ο κύριο Τόρβαλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είχα πει και την προηγούμενη φορά. Να μην αισθάνομαι και σαν παπαγάλος. Σύντομα μόνο θα ήθελα να πω τα κύρια σημεία. Ανησυχούμε όλοι μήπως το γενικό κόστος του προϋπολογισμού ήτρε κινδυνεύει να ε, κατασπαράξει εν τέλει τα υπόλοιπα κονδύλια. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Θα μπορούσαμε να ε, ορίσουμε αυστηρά όρια για το ίτερ με δική του γραμμή του προϋπολογισμού μέσα στα γενικά όρια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, σαν λύση, θα ήταν να αυξήσουμε το ανώτατο του όριο και, με αυτό το, και να το προσδιορίσουμε επίσης, πάλι να θέσουμε δηλαδή πολύ αυστηρά όρια, αυξάνοντας όμως το όριο, ε, για να μην καταναλώσει κονδύλια από αλλού. Τώρα αυτό έχει διαφορε... συνιστά ε, δύο διαφορετικές λύσεις, γιατί αν μείνει μέσα στο α1 θα παρακολουθήσει τον πληθωρισμό και οπωσδήποτε θα απορροφήσει κονδύλια από άλλους σπόρους. Με την, ε, την αριθμική προσαρμογή των προμηθειών στο όλο έργο θα φάει σιγά σιγά τα άλλα κονδύλια. Ανεξαρτήτως τι θα κάνουμε μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η άλλη δυνατότητα να τα αφήσουμε, αυξάνοντας όμως τα ανώτατα του όρια, θα οδηγήσει σε άλλα προβλήματα διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν οι κυβερνήσεις. Είναι πιθανό δηλαδή να πούνε, α, δεν τα δίνουμε τα λεφτά. Αν το βγάλουμε δηλαδή έξω από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν ξέρουμε τι μοίρα θα έχει. Άρα είναι τόσο περίπλοκο όσο και ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Πώς θα το, ε, πού θα το εντάξουμε, πώς θα το διαφυλάξουμε. Και βέβαια πρέπει και την απόφαση να τη λάβουμε ανάλογα με τα δύο αυτά μελήματα. Είμαι διτεθειμένος να ακούσω κάθε πρόταση. Ε, περιμένω να δω τις απόψεις των συναδέλφων της Επιτροπής πριν να υποβάλω τη δική μου ερμηνεία ή πρόταση για το πώς θα το χειριστούμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Γιούτα Χάουκ. Ζήτησε τον καφέ mm-hmm. και τον λόγο. Ευχαριστώ. Είχαμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό και στην προηγούμενη επιτροπή. Προηγούμενη συνεδρία τη επιτροπή μα. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε ένα περιθώριο ακόμη να το αναλογιστούμε και πάλι. Δεν υπάρχει λόγο να αποφασίσουμε αμέσω. Αν και συμφωνούσαμε με όσα είχε πει ο κύριο Στόλβαξ πλήρω. Κατόπιν ορίμου σκέψεως λοιπόν θα πρότεινα εμείς ως Επιτροπή των Προϋπολογισμών να ακολουθήσουμε την πρόταση της Επιτροπής και να βγάλουμε το ΙΤΕΡ από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πλήρως. Έξω από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, από τον Α. Την τελευταία δεκαετία διαπιστώσαμε ότι όταν το ΙΤΕΡ βρίσκεται μέσα στο 1α, απορρόψει συνέχεια όλο και περισσότερα χρήματα και κάθε χρόνο είχαμε την αγωνία που θα βρούμε τα λεφτά γιατί βεβαίως ε, τα περισσότερα χρήματα έτσι άλλωστε επιδιώκουμε και όλα αφορούν ε, το πρόγραμμα έρευνας και όπως υπόθηκε ήδη πάντοτε το πρόγραμμα έρευνας ε, σιγά σιγά μειώνεται λόγω της απορρόφησης των κονδυλίων από το Twitter. Και πρέπει να το κάνουμε γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν καταφέρουμε να ρυθμίσουμε, να διαπραγματευτούμε και να ρυθμίσουμε με το Συμβούλιο θέματα έτσι ώστε να έχουμε και μακροπρόθεσμα αρκετά κονδύλια για το Ίτερ, Αυτά τα οποία έχει προτείνει ήδη τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ίτερ είναι πολύ λίγα κονδύλια, είναι πολύ λίγα όχι γιατί λέμε εμείς α, πρέπει να δώσουμε πιο πολλά λεφτά στο ίτερ έτσι, αλλά γιατί υπάρχουν ήδη ε, συναυθήσεις διεθνείς συμβάσεις για, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν και ως εκ τούτου τα προτινόμενα για το ίτερ κονδύλια μέχρι το 2020 δεν πρόκειται να αρκέσουν. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να κάνουμε τη ζημιά στο 1α και αν δεν θέλουμε να αποκλίνουμε ακόμη περισσότερο από την ε, δεδηλωμένη βούλησή μας για ανταγωνιστικότητα, για καιροτομία, για θέσεις εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είναι καλό να βγάλουμε το ίτερ από την ε, κατηγορία 1α. Ευχαριστώ πολύ, Ιούτα. Άλλες παρατηρήσεις για τον εισηγητή. Σερβατόφ. Εξ ονόματος του σκιωδός εισηγητή Καρβάλιο έχω κάποια πράγματα να σας πω γιατί δεν μπορούσε να είναι παρόν ως σκιώδης εισηγητής για το ITER. Καταρχήν το ITER είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο και τα Πανεπιστήμια και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιστημονική έρευνα. Κατά δεύτερο λόγο συμφωνεί ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου συμφωνούν με την πρόταση της Κομισιόν για 700 εκατομμύρια ευρώ για το περίοδο 2014 μέχρι 2020. Επίσης θεωρεί ότι, ε, ότι θα πρέπει να γίνει διάμεση έκθεση για το PDP έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό ενώ ταυτόχρονα θα χρηματοδοτηθεί η χρηματοδότηση και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων από πιθανές μεταφορές υπέρ του Ήτερ. Ε, ε, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο θα υπάρξουν μελλοντικέ διαπραγματεύσει για το ΠΔΠ. Ε, σε σχέση τώρα με το, διαχείριση του προγράμματος ITER, ε, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική διαχείριση ώστε να αποφευχθεί κόστος, μάλλον υπερβολικό κόστος στο μέλλον. Τέλος, ε, θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο εποπτεύοντας και ελέγχοντας το κονδύλι του προγράμματος. Αυτή είναι η γνώμη του σκιώδου, του σκιώδου σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θέλω να πω ότι και εγώ συμφωνώ ότι το πρόγραμμα ITER θα πρέπει να είναι εκτός του πολιτού δημοσιονομικού προγραμμάτου καθώς ε, όπως είχε συμφωνηθεί και στην συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 7 και 8 ε, ε, εάν παραμείνει μάλλον όπως είχε συμφωνηθεί από το Συμβούλιο 7 και 8 Φεβρουαρίου κινδυνεύουμε προγράμματα όπως το ίτερ να απορροφηθούν από κάποιο άλλο τίτλο, κάποια άλλη κατηγορία του πολιετούς προγράμματος. Εάν ε, θέλουμε ο Ευρωπαϊκό Υπολογισμό να δημιουργήσει θέσει απασχόληση και να διευρύνει ε, τα ερευνητικά προγράμματα ώστε να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, πιστεύω πω είναι προτιμότερο και θα ήταν πολύ καλύτερο το ίτερ να μείνει εκτό του PVP. Merci bien. Ευχαριστώ. Άλλες παρατηρήσεις. Γκέραν. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα απλά να συνεχίσω με βάση αυτά που είπε η Γιούτα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και συμφωνώ μαζί τη, ε, απλά ήθελα να δω τα νούμερα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ότι το ΙΤΕΡ όντω έχει πολύ λίγα χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι διεθνεί μα ε, δεσμεύσει και υποχρεώσει. Ε, αυτό σημαίνει πως ήδη από το 14 το ίτερ θα είναι στην κατηγορία 1α. Ε, μπορεί η Κομισιό να το επαληθεύσει αυτό, ότι τα νούμερα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι υπερβολικά χαμηλά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς μας συμφωνίες για το ίτερ. Γιατί ε, σε τέτοια περίπτωση από την πρώτη μέρα θα έχουμε τεράστιες δυσκολίες στην κατηγορία 1α. Μπορείτε να το επαληθεύσετε από, πλε... από πλευράς Κομισιόν υπάρχει κάποιος εδώ που να είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται όχι. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε ένα πρόγραμμα. Είναι θεμελιώδη αυτή η ερώτηση, ε, αυτό το θέμα. Non, il n'y a pas d'autre demande de parole pour l'instant. C'est une question fondamentale parce que ε, Είναι θεμελιώδες το ερώτημα, γιατί έχουμε δύο ανησυχίες για αυτό το θέμα, θα το θυμάστε. Εδώ και πολλούς μήνες δουλεύουμε για το σχέδιο του πολιετούς πλαισίου και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριτές μας ε, χρειάζεται ένα γενικό προσανατολισμό πρώτη προβληματισμό είναι να είμαστε βέβαιοι ότι η χρηματοδότηση αυτών των μακροχρόνιων προσχεδίων, ε, το ΙΤΕΡ, έχουμε και το Γαλιλαίο και το GMS, ε, που είναι στην ίδια κατηγορία και πρέπει να εξασφαλιστούν. Και ιδιαίτερα ένα σχέδιο, όπως, ένα πρόγραμμα όπως το ΙΤΕΡ, το οποίο σημαίνει πολιτικές και νομικές διεθνείς δεσμεύσεις, όπως είπε και ο Γκέραν Φέρμα. Ταυτόχρονα επιθυμούμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να αποφύγουμε οι υπερβάσεις κόστος που είναι κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτες σε τέτοια καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα να χρηματοδοτηθούν εις βάρος άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως γνωρίζοντας μάλιστα ότι σε περίπτωση του είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο όμως είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των ερευνητικών μας εργαστηρίων, μάλλον σε άλλους τομείς θα πρέπει να δώσουμε μέσα. Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα ε, χρονικής κλιμάκωσης, μάλλον ε, κατανομής. Και ταυτόχρονα θέλουμε και να διατηρήσουμε την αγκαιριότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και είναι ένα σημείο στο οποίο θα επιμείνουμε για τις διαπραγματεύσεις του πολιετούς πλαισίου. Ο καλύτερος συνδυασμός ανάμεσα σε αυτές τις ανησυχίες της πλέον είναι να βάλουμε το ίτερ και ενδεχομένως ένα-δυο άλλα προγράμματα εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου. Αντίθετα, μήπως πρέπει να μπουν στον προπολογισμό αλλά με κάποιες εγγυήσεις. Και εδώ στρεφόμαστε λοιπόν και σε αυτό το ερώτημα που θέτει ο Γκέραν Φέρμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητή μα θα πρέπει να έχει απαντήσει πριν να μα κάνει συγκεκριμένε προτάσει. Κάποιο άλλο. Όχι. Ωραία. Να θυμίσω ότι για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 6 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε στις 26 γιατί πρέπει η Ήτρη να ψηφίσει πολύ γρήγορα γιατί ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην καρδιά των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο σημείο 3 που είναι το σημείο της κατάστασης πρόοδου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δυστυχώς ο Μπέγκε δεν μπόρεσε να είναι παρόν, αλλά έχουμε εδώ τους άλλους μας εισηγητές. Όλοι έχουμε παρακολουθήσει καθημερινά τις εξελίξεις. Επίσης και σε σχέση με την προηγούμενη μας συνεδρίαση θα πρέπει να, να συνειδητοποιήσουμε ότι θελήσαμε και μάλλον ε, κάναμε μια ομάδα επαφής με τον πρόεδρο Σούλτς για να ενημερώνουμε για την κατάσταση, τις εξελίξεις, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφοροι, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε και για να προετοιμάσουμε στη συνέχεια τη διαδικασία στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου. Διαπίστωσα λοιπόν Μάλλον πήγα στο Δουβλίνο ΔΕ για δύο μέρες στις αρχές εβδομάδας με την ευκαιρία της ετήσιας διάσκεψης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οικονομίας και Προπολογισμών, ε, δηλαδή Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι μπόρεσα να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της Ιρλανδίας, ε, ε, της κυβέρνησης, που είναι και υπουργό εξωτερικών, που κατά διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας θα προεδρεύει του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και θα είναι άρα ο συνομιλητής μας όσον αφορά το πολιετές πλαίσιο, ε, συνομιλητής λοιπόν του Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να ε, συναντήσω τέτα τέτ τον πρόεδρο Φανρομπόη που ήθελε να μου εξηγήσει εις βάθος και λεπτομερώς πώς πήγαν τα πράγματα στο Συμβούλιο της 8ης ε, Φεβρουαρίου και να του πω εγώ που βρίσκονταν από πολιτική σκοπιά στα πράγματα στο Κοινοβούλιο. Και είχα έτσι την ευκαιρία Απέναντι στους δύο κύριους ε, ε, αρχηγούς των διαπραγματεύσεων, να επαναλάβω και να θυμίσω αυτό που πάμε από την πρώτη μέρα, αλλά το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχε ακουστεί. Δεν είχε γίνει κατανοητό. Ότι από την πρώτη 12 2009 ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και ότι αυτή η συνθήκη δεν έχει αλλάξει τη διαδικασία υιοθέτηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς έχουμε την ίδια διαδικασία. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα το οποίο η θέση υιοθετείται unblock ή απορρίπτεται unblock με μια μοναδική ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου με πλειοψηφία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Όμως η συνθήκη της Λισαβόνας Κοινοβούλιο την αρμοδιότητα την πλήρη αρμοδιότητα την οποία έχει από με το Συμβούλιο των Υπουργών σε θέματα συναπόφασης, σε θέματα λοιπόν νομοθεσίας, νομοθετικά για τις πολιτικές δηλαδή που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για δημοσιονομικά θέματα όσον αφορά το σκέλος των ετησίων ταπανών ε, για τη συναπόφαση και η θελημένα αγνοώντας αυτή την ε, σοβαρή νομική αλλαγή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προχώρησε όπως και η προκάτοχή του, συμφωνώντας για τις οροφές δαπανών στις μεγάλες κατηγορίες δαπανών, εκεί συμφωνούμε είναι λογικό, είναι η συνθήκη, αλλά και μπαίνοντας σε ένα βαθμό λεπτομέρειες όσον αφορά την κατανομή αυτών των δαπανών και κυρίως τον τρόπο κατανομής ανα υποκατηγορία και εμέσως ή και εμέσως αναχώρα. Και μάλιστα σε τέτοιο, με τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας που σημαίνει πως το Συμβούλιο εκ των προτέρων παίρνει θέση για θέματα και επιλογές και αποφάσεις και κείμενα τα οποία πλέον 100% εμπίπτουν στη διαδικασία συναπόφασης. Και αυτό είναι πρόβλημα. Σε σχέση με τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Έχουμε δύο θέματα αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πολιτικής φύσης για το επίπεδο του προϋπολογισμού. Αυτή η αντιπαράθεση υπήρχε ανέκαθεν, αλλά αυτή τη φορά έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί για πρώτη φορά αυτό που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μείωση του προϋπολογισμού για τα επόμενα 7 χρόνια. Παλιότερα η αντιπαράθεση αφορούσε το μέγεθος της αύξησης. Τώρα πρόκειται για μείωση. Κλασική πολιτική αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό. Υπάρχει και όμως και θεσμικό θέμα. Σήμερα το πρωί συμμετείχα στην συνεδρίαση των ε, Προέδρων των ε, Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου υπό την Προεδρία του Προέδρου Λένε με όλους τους συναδέλφους μας και ο πρόεδρος της ΑΦΚΟ και της Ζούρι το επιβεβαίωσαν ότι τα συμπεράσματα 48 σελίδων που προέκυψαν στις 8 Φεβρουαρίου από το Συμβούλιο ήταν στην ουσία πραξικόπημα. Πραξικόπημα. Το Συμβούλιο από μόνο του ανέλαβε υπεραρμοδιότητες, υπερεξουσίες δημοσιονομικές και νομοθετικές. Γιατί για τον προϋπολογισμό μπορεί να ορίσει υπό την ε, επιφύλαξη έγκριση του Κοινοβουλίου ανώτατα όρια. Αλλά από τη στιγμή όπου τα ανώτατα όρια κατεβαίνουν και κατεβαίνουν μάλιστα τόσο πολύ όσο στην πράξη χρόνο με το χρόνο ο πραγματικός προϋπολογισμός θα είναι καταδικασμένος να βρίσκεται πάντα στην οροφή και δεν θα μπορούμε δηλαδή να τον τροποποιήσουμε παρά την οροφή. Άρα το περιθώριο λιγμού στον ετήσιο προπολογισμό του Κοινοβουλίου περιορίζεται στο μηδέν θα έχετε ίσως υπολογίσει δε ότι επί τη βάση των ανώτατων ορίων των πλαφών που προτείνει το Συμβούλιο για το 2014, γιατί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχει ένα γενικό ε, πλαφόν, 160 εκατομμύρια υποχρεώσεων και μετά υπάρχει η κατανομή ένα χρόνο. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για του χρόνου, οι υποχρεώσεις, ε, το πλαφόν των υποχρεώσεων για τον επόμενο χρόνο θα είναι 12 δις κάτω από τις ε, υποχρεώσεις του πραγματικού προϋπολογισμού του 2013, του πραγματικού όχι της ε, οροφής και για τις πιστώσεις πληρωμών 10 δις λιγότερα. Ωραία τα νέα για την, για εκλογική χρονιά 2014. Δηλαδή 10 δις λιγότερα θα δώσουμε έτσι. Αυτό είναι το σύμφωνο της ανάπτυξης ε, που ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, με ε, την Πανοκρουσίως, ότι δηλαδή θα δίναν ένα σωρό δις για την στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. κόπημα λοιπόν για τις εξουσίες σε επίπεδο προϋπολογισμού και πραξιπόκτημα σε επίπεδο νομοθετικής εξουσίας, γιατί η νομική έρευνα που έγινε από τις νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την οριοθέτηση μεταξύ των θεμάτων που είναι θέματα προϋπολογισμού και αυτών που είναι θέματα νομοθετικά που υπόκεινται στη συναπόφαση δείχνουν ότι τα δύο τρίτα ή τα τρία τέταρτα του κειμένου είναι για θέματα τα δύο τρίτα τα τρία των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορούν θέματα τα οποία είναι συναπόφαση. Το παρουσίασα αυτό στην Κυπριακή Προεδρία. Του ε, έδειξα το κείμενο το οποίο λεγόταν τότε κοιτίων διαπραγμάτευση και όπου υπήρχαν υπογραμμισμένα με χρώματα τμήματα τα οποία υπέκυντο στην ε, συναπόφαση κάναμε το ίδιο πράγμα για το, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το ποσοστό είναι αντίστοιχο. Πρόκειται λοιπόν για ένα πραξικόπημα το οποίο θέλησε να κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να το επιβάλλει σε εμάς, χωρίς αυτό βέβαια να φαίνεται οφθαλμοφανές καταρχήν, γιατί έκανε ακριβώ το ίδιο που κάνανε τα προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Η ανάλυση λοιπόν που κάναμε εδώ ως Επιτροπή Προϋπολογισμών πολλές φορές που την κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα όταν γίνεται το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2011 μετά <clears throat> τα, στα επερχόμενα συμβούλια. Ο, τα θέματα αυτά που έχει τονίσει ο πρόεδρος Σούλτς ενώπιον των διαδοχικών προεδριών και της Προεδρίας Συμβουλίου, ίσως τώρα για πρώτη φορά αρχίζουν όλα αυτά να εισακούονται. Και για πρώτη φορά υπάρχει και κάποια ανησυχία από την πλευρά του Συμβουλίου για τη συνέχεια που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Γνωρίζοντας ότι και μιλήσαμε για το θέμα αυτό με όλους τους συναδέλφους από τις ε, επιμέρους επιτροπές και στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο στόχος μας είναι να διοργανώσουμε τη διαπραγμάτευση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν δύο πτυχές, μια διτή λοιπόν διαπραγμάτευση από τη μία πλευρά για τα θέματα του προϋπολογισμού και κατά τα άλλα για τα νομοθετικά θέματα. Για τα νομοθετικά θέματα τώρα, Τη νομοθετική πτυχή. Τα ανέφερα αυτά στον κύριο Φαν Ρομπέι, τα ανέφερα στον ε, αντιπρόεδρο της Ιρλανδικής Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γκίλμορ. Μα είπαν για όλα αυτά δεν μιλήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν είναι θέματα συναπόφασης, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει πλήρως τις εξουσίες του. Επομένως, εγώ παρότρινα τους φίλους μου από τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου να μην αυτολογοκριθούν αλλά να ασκήσουν πλήρως τις εξουσίες τους. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας το ότι από τη στιγμή στις πιο πολυδάπανες κατά κάποιο τρόπο πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικά ταμεία, γεωργική πολιτική, μεταφορές, έρευνα επίσης, από τη στιγμή που οι επιτροπές θα ασκήσουν το δικαίωμα των τροπολογιών τους. Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία είχε θεσπίσει το Συμβούλιο και τα οποία θα πρέπει να τροποποιηθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν ποσοστά τα οποία θα αλλάξουν. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι κάποιος δικαιούχος ενός προγράμματος ή όχι. Υπάρχει κατάλογος αποδεκτών για κάθε πρόγραμμα. Όλα αυτά θα αλλάξουν. <clears throat> και ιδίως δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τις επιμέρους επιτροπές. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσει ώστε τα ποσά τα οποία έχουν καθοριστεί ανά χώρα ή ανά περιφέρεια θα πρέπει να δικαιολογούνται επί τη βάση κριτηρίων όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικών στις εθνικές μας νομοθεσίες η παράδοση θέλει, αν θέλουμε να υπάρξει μια πολιτική, μια επιδότηση σε ένα οικονομικό κοινωνικό φορέα, σε μια τοπική περιφερειακή οντότητα, θα πρέπει πάντα να εξευρεθεί μια νομική βάση για κάτι τέτοιο. Βάση του κοινωνικού συμφέροντος, του οικονομικού συμφέροντος, του γενικού συμφέροντος αυτή η κατάσταση. Αν υπάρχουν ε, ρυθμίσεις κατά αποκοπή, αν υπάρχει επισφαλής κατάσταση του δικαιούχου, να ληφθεί υπόψη και όλα αυτά. Αυτό μπορεί να ισχύει εν μέρει για τα κριτήρια που προτείνει το Συμβούλιο, τα οποία μπορούμε να τα διαμφισβητήσουμε και να τα αλλάξουμε. Αλλά η γραμματεία κάνει και ένα κατάλογο που σας τον διένυμε. Είναι ο κατάλογος δώρων, οι μπουναμάδες. Είναι αυτά τα ποσά τα οποία δίδονται σε ορισμένες χώρες ή σε ορισμένες περιφέρειες είτε από το ένα ταμείο είτε από το άλλο ταμείο χωρίς όμως να υπάρχει περαιτέρω διευκρίνηση ούτε για τους αποχρόντες λόγους για τους οποίους επελέγησαν αυτές οι χώρες οι περιφέρειες ούτε για το λόγο που επελέγει το ποσό ούτε για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Το καταλαβαίνουμε <clears throat> γιατί το κάνει αυτό. Πάντα αυτό γίνεται, δεν το επικρίνουμε αυτό καθεαυτό. Καθένα με τα προβλήματά τους. Αλλά τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνα. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να μπουν σε μια ανοιχτή δημοκρατική δικαιολογήσιμη διαδικασία όπου είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι με το Συμβούλιο ενώπιον των πολιτών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούμε να αιτιολογήσουμε και να υποστηρίξουμε ενώπιον των πολιτών. Και αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε ένα αποτέλεσμα για τα θέματα αυτά πριν από τις ευρωεκλογέ που θα υποβληθούμε στην κρίση των εκλογέων μας. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω στους εκλογείς μου έγινε μια συζήτηση, ο Α ήθελε αυτό, ο Β ήθελε εκείνο και αποφασίστηκε το τάδε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι απλώς έλαβα γνώση των αποτελεσμάτων και δεν έχω κάνει τίποτα για να τα αντικρούσω. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αλλάζει το σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ξεκινήσαμε από ένα σύστημα το οποίο ήταν διακυβερνητικό. Σιγά σιγά γίνεται ενωσιακότερο. Θεωρούμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ένα ορόσημο αποφασιστικό για αυτό το σύστημα για να γίνει σχεδόν πλήρως δημοκρατικό. Όσο πιο δημοκρατικό γινόταν, όσο πιο διάφανο, όσο πιο υπεύθυνο έναντι των πολιτών μας. Λοιπόν, θα πρέπει να οργανώσουμε επομένω τη διπλή αυτή διαπραγμάτευση και το Συμβούλιο από τη δική του πλευρά θα πρέπει και αυτό να ξεκινήσει τις διπλές αυτές διαπραγματεύσεις για το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε δύο άγνωστους χ σε αυτή την υπόθεση. Πρώτα το χρονοδιάγραμμα. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου, όπως γνωρίζετε, εμείς θα προετοιμαστούμε να καταθέσουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα δώσει απάντηση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην επόμενη ε, Σύνοδο στις 13 Μαρτίου καταρχήν. Και επομένω οι εισηγητέ, οι ομάδε εργάζονται για τα θέματα αυτά για να συγκροτηθεί αυτό το ψήφισμα. Έγιναν πολλέ συναντήσει χθε για όλα αυτά. Δεν πρόκειται να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα ποια είναι τα σχέδια ψηφίσματο τα οποία θα υποβληθούν από του εισηγητέ. Και τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ο στόχο του Πρόεδρου Σούλτ, όπω και τον εξήγησε στην ομάδα επαφή, είναι όπως εξάλλου το αναφέρει σήμερα στον Έντα Κέννη στο Λουβλίνο και στον Πρώτο Παρόσο, είναι να γίνουν τα πράγματα τα οποία είναι τα απαραίτητα, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις από τις 13 Μαρτίου το βράδυ. Το Κοινοβούλιο δεν είναι ικανοποιημένο από τα, από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, θα το εκφράσει αυτό στις 13 Μαρτίου και συνέχεια είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί από τι 10 Μαρτίου. Από την πλευρά του Συμβουλίου. Ε, εκεί είναι τα πιο διασκέστικα πράγματα γιατί το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο. Το Συμβούλιο θα είναι στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τον Προπολογισμό και για την Περιφερειακή Πολιτική. Εκείνη οι αρμοδιότητε του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και μετά το Συμβουλίο Υπουργών Γεωργία για τα αγροτικά θέματα κτλ. Το γενικό πλαίσιο θα καθοριστεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνεδριάζει τη Δευτέρα, αλλά δεν έχει το θέμα αυτό στη μέση διάταξή του. Δεν είναι έτοιμη τεχνικά, δεν έχει γίνει η διαπεξεργασία, πολιτική επεξεργασία, δεν ξέρω τι φταίει, δεν είναι έτοιμη. Τον Απρίλιο λοιπόν και μόνο το Συμβούλιο θα εγκρίνει την εντολή διαπραγμάτευση από την πλευρά τη Ιρλανδικής Προεδρία. 22 Απριλίου θα γίνει αυτό. Δύο μήνες λοιπόν έχουμε μπροστά μα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και νωρίτερα. Πρώτο ερώτημα. Ποιο θα είναι το πραγματικό χρονοδιάγραμμα. Ίσως θα γυρίσει ο Μάρτιν Σούλτς από το Δουβλίνο με έχοντας νέες και διαφορετικές πληροφορίες. Εγώ σας λέω αυτά που ξέρουμε τώρα. Δεύτερο ερώτημα ποιος θα έχει την ευθύνη και με ποιο τρόπο για να μετατρέψει σε να επενδύσει με νομικό ένδυμα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές πράξεις. Μπορούμε να πούμε μια μεριά είναι νομοθετικό θέμα, την ε, πρωτοβουλία έχει η Κομισιόν, εναπόκειται στην Κομισιόν είτε στο να ξαναγράψει τους κανονισμούς για τα Ταμεία Συνοχής, για το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να παρουσιάσει κάποια ε, άρθρα στους κανονισμούς αυτούς με νέα μορφή. Αν γίνει κάτι τέτοιο όμως, τότε θα πρέπει η Κομισιόν να αποδεχθεί όλα αυτά τα οποία είπε το Συμβούλιο. Αυτό είναι και ευθύνη της Κομισιόν. Ο Ντομινίκ Ρικέ θα σας σχολιάσει αυτό το θέμα. Εγώ σας τα λέω τα πράγματα όπως είναι τώρα, όπως τα γνωρίζω εγώ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι όλη η πραγματικότητα. Ή αλλιώς θα θεωρηθεί ότι εφόσον είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο έχει ξεκίνησει αυτή η διαδικασία είναι οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου, η γραμματεία του Συμβουλίου που θα πρέπει να υλοποιήσει σε νομικό επίπεδο τις αποφάσεις αυτές <clears throat> και αυτές θα είναι και οι εντολές διαπραγμάτευσης για την πλευρά του Συμβουλίου. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια να επιφυλάσσεται του δικαιώματο να κάνει νέες προτάσεις στη συνέχεια εν ώψη του τρόπου με τον οποίο η νέα θέση του Συμβουλίου Υπουργών θα γίνει θα τύχει αντιμετώπιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από του διαπραγματευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εν ώψη των τροπολογιών που θα διατυπώσει η πλευρά του Κοινοβουλίου. Αυτό το σημείο λοιπόν δεν είχε ακόμα ξεκαθαριστεί σήμερα το πρωί. Μίλησα χθε με τον πρόεδρο Μπαρόσο, αλλά δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Και όσο δεν έχουμε περαιτέρω διευκρινίσει για το ποιο θα κάνει τι, ως προς το what next, ως προς το who's in charge, ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος για το επόμενο βήμα και με ποια μορφή. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από ό,τι μας επιτρέπουν οι άλλοι εταίροι. Αυτά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτές είναι οι πιο φρέσκες πληροφορίες που έχω. Θέλουν οι συγητές να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν αυτά που είπα πριν δώσω το λόγο στον Ντομινίκ και στους άλλους συναδέλφους. Υπάρχει κάποιος άλλος? Ο Ήβο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Έχω και μια πίεση χρόνου λόγω του αεροπλάνου που πρέπει να προλάβω, αλλά θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία ακόμη, γιατί έχουμε ήδη την, ε, ξεκινήσει την επεξεργασία του ψηφίσματος με τον κύριο Μπογκέ. Ελπίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα διανεμηθεί, εφόσον το οριστικοποιήσουμε. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι πρέπει να είναι σαφές πως δίνουμε εντολή για διαπραγμάτευση μέσω του ψηφίσματος. Και πρέπει να είναι σαφής η εντολή για διαπραγμάτευση δεν αποφασίζουμε εάν θέλουμε ή δεν θέλουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτό θα το κρίνουμε μόνο όταν ε, καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις και κρίνουμε αν είναι επιτυχής ή όχι. Το ψήφισμα λοιπόν αφορά την διαπραγμάτευση. Τα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση, για τη μορφή που έχουν, δεν μπορούν να εγκριθούν. Δηλαδή, καθιστώ σαφέ ότι δεν υπερψηφίζουμε ούτε καταψηφίζουμε τα συμπεράσματα. Ακούω κάποιου συναδέλφου που φαίνεται να αντιλαμβάνονται πω τώρα ψηφίζουμε, υπερψηφίζουμε, καταψηφίζουμε. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Απλώ δίνουμε εντολή για διαπραγμάτευση. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, στη διαπραγμάτευση πρέπει να δώσουμε σαφή εντολή και να πούμε ότι χωρί αυτέ τι διαπραγματεύσει δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν τα συμπεράσματα. Ο πρόεδρο, πολύ σημαντική διευκρίνηση και θα θυμάστε ασφαλώς ότι νομικά για το πολίτες νομικό πλαίσιο το ΣΥΠΗΝ. Υπάρχουν τρία κείμενα. Ένα από αυτά είναι μόνο στην διαβούλευση και αφορά την απόφαση για του ίδιου πόρου. Τα δύο σημαντικά κείμενα είναι ο κανονισμό πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου με τον πίνακα και τα αριθμητικά στοιχεία ανακατηγορία και αναέτο και η διοργανική συμφωνία που συνιστά τον τρόπο λειτουργία ή εφαρμογή του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Και εκεί μέσα είναι η ευελιξία, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, η παρακολούθηση στι πολιτικέ τη χρηματοδότηση, η εξέλιξη τη δημοσιονομική λειτουργία. Αυτά τα δύο λοιπόν τελευταία κείμενα ε, ακολουθούν ίσως ελαφρώς διαφορετικές μεταξύ τους ε, διαδικασίες, αλλά πρακτικά πρόκειται για μια ψηφοφορία on block, υπέρ κατά. Αυτή όμως ψηφοφορία on block, όπως είπε ο Βάιλο, μόνο στο τέλος της διαδικασίας θα λάβει χώρα, όταν δηλαδή θα έχουμε διαπραγματευτεί το περιεχόμενο. Οι εισηγητές μας καταρτίζουν ένα σχέδιο ψηφίσματος, πολύ σημαντικό, που θα αποτελέσει την εντολή διαπραγμάτευσης, που θα δώσει την απάντησή μας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή θα πούμε εμείς ότι στο, ε, στα συμπεράσματά σας υπάρχουν πράγματα που δεν μας ικανοποιούν, που δεν δεχόμαστε και ορίστε τι προσκοπεύουμε να δεχθούμε. Άρα, η έγκριση του ψηφίσματος αυτού δεν συνιστά οριστική απάντηση εκ μέρους του Κοινοβουλίου και δεν έχει στόχο να κλείσει τη διαπραγμάτευση, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέψει την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Ε, ξέρω, το συστήσαν όλες οι ομάδες, θα το ξανασυζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την ε, σύνοδο στο Στρασβούργο θα το έχουμε το θέμα αυτό. Αλλά όποιος έχει εμπειρία από τη διαπραγμάτευση ξέρουν ότι είναι μια πολύ λεπτή τέχνη, η τέχνη της διαπραγμάτευσης. Και ότι συνιστά ένα έργο μακρόπνο. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δόθηκε η εντύπωση ότι στις 8 Φεβρουαρίου ή άντε το πολύ στις 9 εκρίθησαν τα πάντα. Γιατί θαύμα θαυμάτων, συμφώνησε το Συμβούλιο, κλείσαν όλα τα θέματα κτλ. Στη συνέχεια και χάρη σε μια κοινή αντίδραση προέδρων ομάδων μέσω ενό ανακοινοθέντους τύπου, ε, τα μέσα μας και ενημέρωση ανακάλυψαν ότι υπάρχει και το κοινοβούλιο και ότι ε, προϋποτίθεται μια διαδικασία ψηφοφορίας με έγκριση από το Κοινοβούλιο. Άρα ότι υφίσταται και κίνδυνος απόρριψη από πλευρά του Κοινοβουλίου. Άρα ε, μετέφεραν στην κοινή γνώμη ότι σε 15 μέρες μέσα θα κρίνει το θέμα το Κοινοβούλιο και θα κλείσει κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα χρειαστεί χρόνος. Γιατί το χρονοδιάγραμμα, επί τη βάση του οποίου εργάζεται η Ιρλανδική Προεδρία, προβλέπει δυνατή τελική απόφαση μέσα στον Ιούνιο, ίσως ακόμη και τον Ιούλιο. Και θα συναντήσω σε λίγο τον ε, Λιθουανό πρεσβευτή, γιατί είναι η επόμενη Προεδρία και θα δούμε. Θα το συζητήσουμε και μαζί του. Άρα λοιπόν, πρέπει πρώτα να αντιληφθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά ε, διαπραγμάτευση και πρέπει και εμείς βέβαια να το αντιληφθούμε και να προετοιμαστούμε για αυτή τη μακρά διαπραγμάτευση γιατί θα υπάρχουν διαφορετικά χρονικά σημεία ε, έντασης ενδεχομένως ε, διακοπής των επαφών, ανάληψης επαφών, επανάληψης επαφών. Υπάρχει όλη αυτή η, το, θεατρικό όλο αυτό που ζούμε κάθε χρόνο σε τελευταία ανάλυση γιατί κάθε περίοδος πρέπει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός ε, μέσα σε μερικές ημέρες ή νύχτες για τον ενιάυσιο, για τον ετήσιο προϋπολογισμό ε, υπάρχει ένταση αλλά σε πιο συμπυκνωμένη μορφή Τώρα θα τη ζήσουμε αυτή την ένταση σε πιο ε, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κύριος ε, Ρικέ έχει, το, λόγο. Καταρχάς, Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση που με απασχολεί πολύ και μετά μια παρατήρηση. Η ερώτηση είναι εξής. Υπάρχει μια γραμμή μεταξύ αυτών που ανήκουν στο πολιτισμο νομικό πλαίσιο και εκείνων που υπάγονται στην νομοθετική ε, βάση, στην νομική βάση. Μια γραμμή δηλαδή που ξεχωρίζει αυτά που ε, ανήκουν, υπάγονται στο πολιτισμο νομικό πλαίσιο και τα άλλα που ε, εντάσσονται στην νομοθετική διαδικασία, νομοθετική βάση. Ξέρετε ότι αυτά τα δεύτερα θέματα έχουν ξεκινήσει να συζητούνται και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη Τρεμερή διάλογο για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο, η νομοθετική βάση, η οποία όμω νομοθετική βάση πολύ συχνά έχει και αριθμητικά στοιχεία, νούμερα δηλαδή, είτε ως επικεφαλίδες είτε πιο χαμηλά στην πυραμίδα της ιεραρχίας, ε, για τα οποία όμως νούμερα θα ήθελα να μάθω τι είδους συνέπειες μπορεί να έχουν σχέση με το πολιτές πλαίσιο και θα δώσω ένα παράδειγμα γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ για το Connecting Europe Facility είμαι συγητής και διαπιστώνω ότι στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προσδορίζεται βεβαίως το κεφάλαιο μέσα στο 1α όπου προσδιορίζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι το Connecting Europe Facility για το οποίο προσδιορίζεται και ένα χρηματικό ποσό Τώρα, στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου μπορεί μια νομοθετική βάση να προβλέψει συγκεκριμένο ποσό 30,2 δις, δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά κατανέμεται σε τρεις ε, κατηγορίες, μεταφορές ή σε τρεις κλάδους, μεταφορές, ενέργεια και επικοινωνία, το Connecting Europe Facility. Εδώ πέρα λοιπόν θέλω να ρωτήσω το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι πού θα φτάσει. Σε ποιο βαθμό λεπτομέρειες θα πάει το Συμβούλιο τελικά. Θα μπορεί να μας πει α, μέχρι εκεί και τα πάντα τα καθορίζουμε εμείς ή μήπως τελικά έχει παρέμβει υπερβολικά στην νομοθετική βάση. Αυτή είναι η απορία μου και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για άλλα θέματα, όχι μόνο για το Connecting Europe Facility. Και επίσης, σε κάτι άλλο που αναφέρατε, Μήπως υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και να τα μετατρέψει σε μια πρόταση νομοθετική επί τη βάση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχω την εντύπωση ότι έχει ήδη δώσει την απάντηση η Επιτροπή λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν. Ε, για τη τελευταία ανάλυση, αν μπορούσε να το πράξει, θα είχε ήδη προτείνει ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εγώ αλλά και οι σκιώδεις θέλουμε να ξέρουμε εάν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο για το 2014 που θα συγκεκριμενοποιεί το MFF ε, θα χρειαστεί οπωσδήποτε τη συμφωνία του Κοινοβουλίου, διότι το MFF δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο εάν εγκριθούν ε, από τα δύο σκέλη του προπολογισμού οι προτάσει. Άρα ούτε σχέδιο δημοσιονομικό, ούτε τροποποίηση νομοθετική βάση μπορεί να γίνει έμεσα έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά θα μπορούσε να παραμείνει σε κάθε σημείο της δημοσιονομικής διαδικασίας. Εγώ προσωπικώς δεν ήθελα να ξέρω πού σταματάει η επέμβαση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, μέχρι, που, μέχρι του πολιτικού βαθμού λεπτομερίας σωστικά μπορεί να επέμβει το ε, πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλιώς τελικά δεν έχει και πάρα πολύ νόημα να συζητάμε με τα επιμέρους συμβούλια των Υπουργών, Υπουργών Μεταφορών προκειμένου ή με άλλα συμβούλια εξειδικευμένα ε, εάν ε, τελικά μπορούν να μας παρακάμψουν και να υποχρεώσουν το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να δεχθούν ε, πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα να δεχθούν. Πού βρίσκεται δηλαδή η κόκκινη γραμμή, ποιο είναι το όριο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει το Συμβούλιο. Δύο παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις. θέλει και άλλο. Κύριε συναδελφέ. Και ξεκινώ από τη δεύτερη. Θεωρώ ότι είναι ορθή η ανάλυση σου. Είναι ορθή η ανάλυση σου. Δεν μπορεί να το πράξει δηλαδή αυτό η Επιτροπή. Και με στηρίζει και στο μεταφέρω αυτό που είδα εγώ για τη χθεσινή μου συζήτηση με τον Παρόσο και τον Ζεζόμ, ότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν, είναι, δεν γνωρίζει, δεν προβλέπει σε ποια βάση θα προετοιμάσει τον προπολογισμό του 2004 και για την κυρία Χολμάιερ και την κυρία Γένσεν, πρακτική συνέπεια αυτού είναι ότι δεν θα είναι σε θέση από 1η Μαΐου να καταθέσει το προσχέδιο του προπολογισμού. 1η Μαΐου μπορεί να μας βάλουν να δουλεύουμε, τόσο πάνω, το πολύ δύο. Ε, θα χρειαστεί να περάσει πιο πολύ χρόνο για να ετοιμάσει το προσχέδιο του προπολογισμού. Μα λέει δηλαδή ότι δεν μπορεί ούτε σχέδιο προπολογισμού να ετοιμάσει επί τη βάση των αρχικών τη προτάσεων και να το υποβάλει στο κοινοβούλιο με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ε, εκφέρει γνώμη το Κοινοβούλιο, άρα θα πρέπει να δείξει μια μεγαλύτερη ε, δημιουργικότητα και φαντασία, εκτός βέβαια και αν προλάβουμε μέσα στον Απρίλιο να καταλήξουμε συμφωνία με το Συμβούλιο, αλλά διαφορετικά θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις η Επιτροπή. Για το πρώτο ερώτημα, πρέπει πρώτα το Κοινοβούλιο να εκφράσει τη δική του ερμηνεία. Και αυτό σημαίνει ε, ανάληψη επαφών με τους ε, προέδρους των εμπλεκομένων επιτροπών και να προσδιορίσουμε τι θέλουμε εμείς ως κοινοβούλιο. Γιατί το λέω αυτό. Διότι έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία ανακατηγορία, υποκατηγορία, που έχει καταγράψει το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του. Αλλά και μετά πρέπει να γίνει η κατανομή των ποσών στη λεπτομέρειά τους. Η λεπτομέρεια λοιπόν αυτή μπορεί να επαφεθεί, μάλλον ε, ε, ουσιαστικά επαφείεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκείνη θα πρέπει να κάνει την πρόταση. Γιατί τη λεπτομερή όμως κατανομή, την ίδια δυσκολία με αυτήν την οποία αναφέρατε μόλις τώρα αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορεί δηλαδή να καταθέσει νέες λεπτομερείς προτάσεις με δεδομένα μόνο τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς την έκκληση του Κοινοβουλίου. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι εμεί, το Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή των Προπολογισμών, θα πρέπει να είμαστε θέση να πούμε ε, δεχόμαστε το ποσό αυτό ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μας δώσει κανένα δύο δισεκατομμύρια παραπάνω το Συμβούλιο, το δεχόμαστε έστω και από εκεί και πέρα να πούμε τώρα πρέπει να πούμε ποιος είναι ο καταμερισμός, πώς μοιράζονται τα ποσά. Και ενδέχεται, ενδέχεται μάλιστα και να το δεχθεί το Συμβούλιο, να πει το Κοινοβούλιο ότι για το Connecting Europe Facility για τις τηλεπικοινωνίες συγκεκριμένα έγιναν υπερβολικά πολλές περικοπές και αντί για ένα δις, αντί να, να χωρίσουμε το ποσό σε 10 φέτες, θα το μοιράσουμε στα δύο μόνο. Αυτό θα ήταν θεμητό πιστεύω από πλευρά του Κοινοβουλίου και δεν θεωρώ ότι μπορεί να ε, προξενήσει αναφανδόν αντίδραση και άρνηση, απόρριψη από το Συμβούλιο. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι εμείς με τις συναρμόδιες επιτροπές ή με τις αρμόδιες επιτροπές ε, θα συμφωνήσουμε. Θα πάρουμε λεφτά από το Ήτρε να τα πάμε στις μεταφορές, τι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να κάνουμε να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτό έλεγα και νωρίτερα, ότι πρέπει να προβλέψουμε δηλαδή πως μια χρονική στιγμή και όταν θα έχουμε πιο πολύ ε, βεβαιότητα σε σχέση με τα αριθμητικά θα πρέπει να κάνουμε την κατανομή των ποσών στα διάφορα έργα. Ο κύριος Τρικέ, ε, ωστόσο θα μπορούσε να προκύψει η πιθανότητα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές βάσεις ε, για τα νομοθετήματα ουσιαστικά του κανονισμού πιο γρήγορα από ό,τι διαπραγματεύσει το πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή να έχουμε τα επιμέρου ποσά και να μην έχουμε το συνολικό ποσό. Και άρα μπορεί να προχωρήσουμε ξεκινώντας από τις νομοθετικές βάσεις και περνώντας μετά σε ένα πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα, θα απορριφθεί. Οπότε θα βρεθούμε σε ένα πραγματικό διέξοδο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το να πούμε πού πάβει ο προσδιορισμός από πλευρά του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου των νομοθετικών βάσεων. Αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει αυτό σε βάση εργασία για την Επιτροπή για την καταναμή των ποσών και για το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν όντω προβλήματα ως προς, τις, ε, ως προς τα συγκεκριμένα ποσά, όπου οι προτάσεις του Συμβουλίου είναι ριζικά διαφορετικές από αυτές της Επιτροπής. Αυτό που ανέφερε στο Connecting Europe Facility οπωσδήποτε και η περιφερειακή ανάπτυξη επίση και κάποια άλλα, όχι πάρα πολλά, αλλά και άλλα ποσά. Κατά τα άλλα θα δούμε οι διαπραγματεύσεις ε, με τι ρυθμούς θα προχωρήσουν. Η Γεωργία, παραδείγματι έχει τη δική της ε, πρικοδότηση με την, ε, με την επιφύλαξη όμως ότι λόγω των καθυστερήσεων στο Συμβούλιο οτιδήποτε έχει να κάνει με ενίσχυση ανά εκτάριο οποιαδήποτε τέτοια βοήθεια μόνο από το 2015 και μετά στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά αυτές ήταν οι λίγες περιπτώσεις. Για τις υπόλοιπες όπως και να έχει θα έχει κοινοποιηθεί η τάξη θα γνωρίζουμε ποια είναι η τάξη μεγέθου, ίσως με κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια διαφορά. Απόκληση. Άρα, εάν πριν από την νομοθετική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία για το Πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορεί να ε, προσδιοριστεί το νομοθετικό τμήμα με ένα ελάχιστο ποσό, να πάρουμε το ελάχιστο απαραίτητο ποσό και αν μετά με τις ε, διαπραγματεύσεις το πολιτισμο συνομικό πλαίσιο εξασφαλίσουμε περισσότερα ποσά, τόσο το καλύτερο, τα συμπληρώνουμε. Πάντως πρέπει να έχουμε ε, παράλληλη εξέλιξη των ε, νομοθετικών διαπραγματεύσεων και των δημοσιονομικών για το πολιτισμό οσυνομικο πλαίσιο. Γνωρίζετε όμω ότι αν το ένα σκέλο προχωρήσει κάπως πιο γρήγορα θα πρέπει να το τραβήξει πίσω και να το καθυστερήσει το άλλο σκέλος. Οτιδήποτε λοιπόν έχει ε, προχωρήσει, εγκριθεί και είναι σε θέση να λειτουργήσει το 2014 πρέπει να ξεκινήσει. Περιφερειακά ταμεία, ε, ταμείο συνοχής, ε, ό,τι προγράμματα υπάρχουν θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς ό,τι προγράμματα είναι έτοιμα, ακόμα και αν δεν ξέρουμε αν το συνολικό ποσό για τη συνοχή θα είναι 50 ε, εκατομμύρια ή 40. 50 δις ή 40 δις. Μπορούμε λοιπόν να προβάλλουμε κάποιες υποθέσεις, το και αν δεν είναι ασφαλής 100% έχουμε μια τάξη μεγέθους ήδη. Αλλά από την άλλη μην καθυστερήσουμε και τόσο ώστε να μην έχουμε, ε, να μην έχουμε καμία ιδέα για το που προχωρούμε, για το που βαίνουμε. Ο κύριος Αλφόνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη στη διαδικασία που έχει ακολουθήσει το Κοινοβούλιο και που επέτρεψε στο Μάρτιν Σούλτς να προβάλλει εξ ονοματός μας τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως και επιθυμούμε οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί τώρα να αποτελέσει συνέχιση αυτής της διαδικασίας και φυσικά ε, δεν θέλουμε να φανεί το κοινοβούλιο σαν ένας μήνος σπουργητιών που διαλύεται με το πρώτο, με την πρώτη, με το πρώτο ασταραπόβροντο, δηλαδή τους ορισμού του Συμβουλίου. Θέλουμε λοιπόν να υιοθετηθεί ένα ψήφισμα, να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, να ε, προχωρήσουμε με βάση αυτό, γιατί ε, εάν έστω κάποια πράγματα μπορεί να φαίνονται αποδεκτά για τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς θεωρούμε ότι για την Ευρώπη, για την Ευρώπη είναι απαράδεκτα. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσδιορίσει ότι είναι αποδεκτό, παραδεκτό για την Ευρώπη και όχι για το κάθε κράτος χωριστά, για το διαλυμένο μήνος. Ε, έχω λοιπόν τρία ζητήματα κυρίως, σύγκληση μεταξύ ε, πιστώσεων, ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, η ευελιξία και η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Τι είδους ευελιξία και τι είδους μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση μπορούμε να συζητούμε όταν έχουμε τέτοια απόκληση μεταξύ ανάληψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Πρόκειται για ε, τέτοιες αποκλίσεις ε, που δεν μας επιτρέπουν να δούμε την πραγματικότητα για αποκλίσεις που ουσιαστικά μας οδηγούν σε μια φενάκη. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό, να καταγγείλουμε τις μεγάλες αποκλίσεις. Το κύριο ζήτημα για μας, για την ομάδα μας, είναι η σύγκληση μεταξύ, απο... μεταξύ ε, πίστασεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών. Ήδη πόροι βεβαίω να είναι γνωστή. και θέλουμε το ψήφισμα να λάβει υπόψη και την προαγωγή των προτεραιοτήτων που έχει προσδορίσει το Κοινοβούλιο. Στη διαπραγματευτική εντολή δηλαδή θέλουμε ιδιαίτερα να ενισχυθεί το κεφάλαιο 1, το κεφάλαιο 4 και ε, η κατηγορία σχετική με την ανάληψη. Γιατί ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Όταν κατά 24% ε, μειώνονται οι πολιτικές εκείνες, η χρηματοδότηση των πολιτικών εκείνων που συνιστούν την ψυχή ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ιδιαίτερα το Εράσμους αλλά και άλλα προγράμματα που προάγουν την ιδέα της Ευρώπης, το να μειώνουμε κατά 24% την προκοδότηση των προγραμμάτων αυτών σημαίνει ότι δεχόμαστε οπισθοδρόμηση ως προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ως προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, σε αυτό πρέπει να αντιδράσει το Κοινοβούλιο και να πει εάν δέχεται την οπισθοδρόμηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δεχθεί και άρα πρέπει να στήσουμε στο 1α, στο 4 ε, σημαντικές ενισχύσεις γιατί δεν αντιλαμβάνομαι παραδείγματι πώς γίνεται να μειώνονται κατά 15-20% αν θυμάμαι σωστά οι πιστώσεις για την εξωτερική πολιτική την ώρα που ζητούμε περισσότερες εντονότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη διεθνή σκηνή και μάλιστα από την πρώτη χρονιά που λέμε ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό με το που διακηρύσουμε την φιλοδοξία αυτή. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερες εξουσίες και χρειάζεται να γνωρίσουμε ότι έχει περισσότερες εξουσίες και δυνατότητες στο Κοινοβούλιο από ότι μερικές φορές φανταζόμαστε και πρέπει να πείσουμε και την κοινή γνώμη ότι υπάρχει αυτή η εξουσία και οι δυνατότητες και θα, πιστεύω, θα βρούμε πιστεύω αν εκδηλώσουμε εμείς τη βούλησή μας και ανταπόκριση στην κοινή γνώμη. Θαυμάσια τα είπατε, σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά, ίσως η υπόλοιπη ομάδα μου δεν με ακούει αυτή τη στιγμή, ελπίζω ότι και η δική μου ομάδα θα πάρει την ίδια θέση μαζί σας. Κατά τη διάρκεια της ε, εποχής πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Παρόσο είχε μια πολύ καλή διατύπωση, είπε. Αυτό που είναι ατυχές με τις επενδύσεις του μέλλοντος, την κατηγορία 1, είναι ότι δεν υπάρχει <clears throat> κάποια εκλογική βάση η οποία να τα υποστηρίζει αυτά τα πράγματα. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μονάχα που υποστηρίζει αυτές τις επενδύσεις του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε, κύριος Διόγκ. Ήθελα να θέσω ένα διαδικαστικό ζήτημα για το ερώτημα του πώς θα λυθεί η απόφαση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ευρέως ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εξετάσει τη χρήση της μυστικής ψηφοφορίας όταν πάρει την τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης των δημοσιονομικών προοπτικών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι αρνητικό για το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω από πού προήλθε αυτή η ιδέα. Η δική μας πολιτική ομάδα χθες εξέφρασε τη στεναρή, τους, ε, τη στεναρή της θέση ότι θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το Κοινοβούλιο δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή τη ε, διαδικασία για μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που έχει να λάβει το Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την επόμενη 7 αιτία. Ελπίζω ότι και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα εκφράσει την αντίρρησή της, την αντίθεσή της σε μια τέτοια πρόπτικη και αυτό θα βοηθήσει να διαλύσει τις παρεξηγήσεις και να σταματήσει τις οικοτολογίες σε σχέση με μια τέτοια διαδικασία. Όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με τη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές προοπτικές. Εδώ άκουσα τον George Lyon με το ε, αριστερό μου αυτή. Το φιλελεύθερο μου αυτή, ενώ το δεξί μου είναι δημοκρατικό. Έχει δίκιο ο George. Τόσο τον μάλλον καθώς αληθεύει δηλαδή αυτό, δεδομένου του ότι προσπαθώ να εξασφαλίσω και πιστεύω θα το εξασφαλίσουμε από το Συμβουλίο και από την Κομισιόν ότι θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια <clears throat> και πλήρης πληροφόρηση για τα πραγματικά στοιχεία που έτυχαν διαπραγματεύσεων και στα οποία κατέληξε το Συμβούλιο. Και αν θεωρούν ότι δεν μπορούν να είναι απόλυτα διάφανοι, το Συμβούλιο και η Κομισιόν, εμείς αντίθετα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε απόλυτα διαφανείς, γιατί επίκυνται οι εκλογές την επόμενη χρονιά ποιο τολμάει να εμφανιστεί ενώπιον των εκλογέων του λέγον ψηφίστε με, είμαι υπεύθυνο άτομο. Και αυτά έκανα στην ε, διάρκεια της θητείας μου, στην πιο σημαντική ψηφοφορία της εντολής μου, που θα αποφάσισε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών και των τρόπων χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών. Μα δεν, σας δεν μπορώ να σας πω ότι ψήφισα γιατί είναι μυστικό. Θα το γράψω στα απομνημονέματά. Η δημοκρατία όμως έχει κάποιες απαιτήσει. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις ευθύνε μας. Αυτό είναι θεμελιώδες. Και αυτή η ιδέα η οποία διατυπώθηκε σε κάποια χρονική στιγμή για να ασκήσει πίεση νομίζω ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος να συμπεριφερθούμε. Είναι ένα όπλο το οποίο θα στραφεί εναντίον μας. Όλα πρέπει να γίνουν με απόλυτη διαφάνεια. Και αυτό με οδηγεί να σας πω αυτό που έπρεπε να σας είχα πει προηγουμένως. Σας έχω στείλει αντίγραφο των ανταλλαγών επιστολών που είχαμε τον πρώτο Πάρασο και τον πρώτο πάει Το ταχυδρομείο αυτό, η ανταλλαγή επιστολών, όπως είπα προηγουμένως, ξεκίνησε από το γεγονός ότι τα σχόλια των 27 πρωτευουσών για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ενθουσιώδη. Ο κάθε ένας πρωθυπουργός έλεγε στη χώρα του ότι ναι, μειώνει, ο προϋπο, μειώνει το προπολογισμό ο πολίτης, αλλά η χώρα του κάτι θρίαβο. Λογικό είναι αυτό. Αλλά το πιο εκπληκτικό, δώσανε και αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με τις επιστροφές που θα παίρνουν οι χώρες τους. Και εγώ αναγκάστηκα να πω χθε ή προχθές στο, στην Προεδρία του Συμβουλίου εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως παρουσιάστηκαν από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ο καθένα στη χώρα του. Γιατί άμα τα προσθέσω όλα αυτά που είπανε, έχουμε ξεπεράσει τα χίλια δισεκατομμύρια. Όχι 960. Και δεν ξέρω ποιο θα τα χρηματοδοτήσει, γιατί όλοι λέγανε ότι έχουν καταφέρει να μειώσουν τι εθνικέ συνεισφορέ. Πολύ όμορφα. Εδώ υπάρχει όμω κάτι το παράδοξο. Εγώ δεν διαφυσβητώ την καλή θέληση και την καλή πίστη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Είναι η πληροφόρησή τους η οποία είναι ελλειπής έχουν κάποιες πληροφορίες που εμείς δεν έχουμε. <clears throat> Θα πρέπει να τις έχουμε λοιπόν και εμείς. Εν κατακλείδη λοιπόν, στα ερωτήματα αυτά λέει ο πρόεδρος της Κομισιόν ότι αυτά τα στοιχεία εγώ δεν τα έχω. Ρωτήστε το Συμβούλιο και ο επικεφαλής του γραφείου του πρόεδρου του Συμβουλίου είπε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, αυτά τα κάνει η Κομισιόν. Οι εισηγητέ μα λοιπόν χρειάζονται να έχουν αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να εργαστούν. Θα πρέπει να ξέρουν ακριβώ ποια είναι τα στοιχεία κατά χώρα, κατά πολιτική, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την απαραίτητη σύγκριση. Εν πάση περιπτώσει, Ζωζ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα δράσει με τρόπο ο οποίος είναι διάφορος, η ΑΙΝΤΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο ακριβώς για αυτό το σημείο. Γιατί έχουν ελεγχθεί ήδη πολλά πράγματα και θα ήθελα να φέρω και ποια είναι η δική μου θέση, η θέση της ομάδας μου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το γεγονός που θεωρούμε εμείς σκανδαλώδες, ότι σε μια χρονική στιγμή που χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, αυτό το οποίο έκανε το Συμβούλιο είναι να περικόψει, να περικόψει και να ξαναπερικόψει. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Θα ήθελα να σταθώ στο ερώτημα το οποίο έθεσε ο πρόεδρος Λαμασούρ. Το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα πραγματικά νούμερα και συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι τη μέρα μετά από το Συμβούλιο ο κάθε επικεφαλής ε, κράτους και κυβέρνησης είπε ότι ναι νικήκαμε στη χώρα του. Με τόσες πολλές νίκες το ερώτημα είναι ποιος έχασε. Τι θα βγει από όλα αυτά. Γιατί φαίνεται ότι όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων διακηρύττουν την νίκη και το θρίαβό τους. Και παρόλα αυτά όλοι ήταν ομόφωνοι με, στην έγκριση της τελικής πρότασης του Συμβουλίου. Για μένα είναι ανησυχητικό το ότι ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβουλίο δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα στοιχεία τα οποία θα μας επέτρεπαν στην πράξη να γνωρίσουμε ποια είναι η πρόταση από την πλευρά του Συμβουλίου για τον προπολογισμό. Δεν είναι παραδεκτό για μας να παραβιάσετε το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά που είναι ένα θεμελιώδες προαπαιτούμενο δημοκρατίας και διαφάνειας. Το να μην ξέρουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά αναχώρα και τα στοιχεία αυτά να μην έχουν παρουσιαστεί στα κράτη μέλη και να υπάρχει μονάχα αυτή η απάντηση που δόθηκε στον πρόεδρο Λαμασόρ. Όχι μόνο θα είναι σε αυτό, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει δεκτό. Γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πλήρους απόφασης και αυτό προϋποθέτει την πλήρη πληροφόρηση του. Αυτό ήθελα λοιπόν να πω. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτό το οποίο έγινε στο Συμβούλιο δεν ήταν μια συνεδρίαση των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένα άθροισμα διμερών ε, συναντήσεων όπου ο πρόεδρος ε, Φαρρομπόι μοίραζε ψίχουλα στις διάφορες χώρες και επειδή όλοι είχαν ψίχουλα στο τέλος κατέληξαν να είναι ευχαριστημένοι χωρίς να κατανοούν ότι με τον τρόπο αυτό αμφισβητούν και υπονομεύουν την, την ε, αλληλεγγύη που είναι απαραίτητη για το ευρωπαϊκό ε, εγχείρημα. Η Ίγκε Γκρέσλερ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Μα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να υπάρχει καινούριο στα οποία ε, συζητάμε και έχουμε και άλλα σημεία στην ημέρηση διάταξη και έχουμε και αεροπλάνα ή πλοία ή τρένα να πάρουμε. Ευχαριστώ, Ίνγερ. Μα το θέμα που συζητάμε δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα, δεν είναι ένα ίσον θέμα. Ο κύριος Κλούγκε και θα περάσουμε στην ημερησία διάταξη. Α, δεν θα μπορέσω να μιλήσω δηλαδή, λέει ο κύριος Κλούτε. Αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα είναι το εξή, ότι παραγωγή χάρη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αυτό το οποίο αναφέρεται στα μέσα ενημέρωση είναι ότι είναι μια θαυμάσια συμβαστική λύση την οποία πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι. Ενώ αυτά τα οποία είπαμε σήμερα δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου έτσι και είναι πολλοί πολίτες οι οποίοι δεν θα δεχτούν αυτή τη συμφωνία άμα δουν τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Πώ λοιπόν είναι το ερώτημα που θα εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτε θα είναι πληροφορημένοι για αυτά τα οποία έχουν πράγματι αποφασιστεί. Είναι πολύ πλοκά όλα αυτά βέβαια, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, πιστεύω, τον τρόπο να εξασφαλίσουμε από τα μέσα ενημέρωση ότι θα προβληθεί η πραγματικότητα. Αυτό το έχουμε συζητήσει και στην ομάδα επαφή. Εγώ νομίζω ότι εφόσον μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό του προπολογισμού, θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα αυτό κατά πόσο οι πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές να είναι μόνο πέντε ετών, δηλαδή να είναι σύγχρονες και παράλληλες με μια κοινοβουλευτική περίοδο ή περίοδο της ε, θητείας της Κομισιόν. Ούτως ή άλλως είναι θεμελιώδες δικαίωμα ενός κοινοβουλίου να αποφασίζει για τα θέματα προπολογισμού και τον έχουμε μια περίοδο ε, προοπτικών που ξεπερνάει τη θητεία ενός κοινοβουλίου, αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα σε επίπεδο δημοκρατίας και θα ήθελα και αυτό να το υπενθυμίσω και να ληφθεί αυτό υπόψη στη συνολική διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Δαμασούρ. Ούτως έχουμε κάνει μια γενική επισκόπηση σε σχέση με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή μόνο τη προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με όλα τα ερωτηματικά τα οποία παραμένουν για την διοργάνωση των διαπραγματεύσεων, για το χρονοδιάγραμμα, για την διαδικασία. Σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 7 που είναι η κοινή παρουσίαση του σχεδίου συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενεδίσεων για τις διαγραφές και τις διαδικασίες του καταμερισμού κινδύνων μέσω των ομολόγων έργου. Project Bonds. Καταρχήν, έχουμε τον διευθυντή, τον γενικό διευθυντή Εκφίν της Κομισιόν, τον κύριο Γιάννη Τόμας, και τον κύριο Νίκ Τζένετ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχετε το λόγο, θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, κύριε Τζενέτ. Εν συντομία μου σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη συμφωνία Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, τράπεζας για την πιλωτική φάση. Ο Δόκτωρ Χόιερ με παρακάλεσε να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του που απουσιάζει σήμερα, όπως ξέρετε. Δυστυχώς ε, νοσή, ασθενή και δεν μπορούσε να έρθει, αλλά ε, ζήτησε συγγνώμη. Πολύ σύντομα λοιπόν. Γνωρίζουν πιστεύω τα μέλη της Επιτροπής σας ποια είναι η λογική πίσω από τα ομόλογα έργου. Η ανάγκη για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσεχή προγραμματική περίοδο, η ανυπαρξία, η ανεπάρκεια καλύτερα του, της δημόσιας χρηματοδότησης, το γεγονός ότι η τραπεζική αγορά που ε, αποτέλεσε την κύρια πηγή χρηματοδότησης των υποδομών τα τελευταία χρόνια ε, είναι λιγότερο προσβάσιμη, καθώς ε, αναζητούν μόχλευση τράπεζες σχέση με το παρελθόν και έτσι για τις υποδομές συμφωνούμε ότι κεφαλουχικές αγορές, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιωτικά συστήματα είναι οι φυσικοί ούτως υπήν χρηματοδότες των μακροπρόθεσμων έργων υποδομών, γιατί με τη σταθερή ροή ρευστότητας μπορούν να αντισταθμίσουν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Επίσης σχεδόν οι πάντες συμφωνούν στο ότι δεν το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό τώρα και δεν συμβαίνει τώρα διότι τα πρωτογενή έργα χρηματοδότησης, τα λεγόμενα Greenfield, δεν βρίσκουν χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν αυτό που αναζητούμε εδώ είναι ένα πολύ εστιασμένο μέσον και αυτό θα αποτελέσουν τα ομόλογα έργου για να καλύψουν τις ανάγκες ε, κάλυψη από ε, επενδυτές ή να, να εγγυηθεί στους εγγυητές ε, το κεφαλαίο τους για τη χρηματοδότηση των έργων. Άρα λοιπόν Στόχος μας είναι να ξανανοίξουμε την κεφαλαιοχική αγορά για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων στις μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Το μέσο το οποίο έχουμε φτιάξει στηρίζεται σε υφιστάμενα μέσα που προσπαθούμε να συνδυάσουμε η Επιτροπή μας με την Τράπεζα και με ε, στήριξη και από μια ε, χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Η Συμφωνία Συνεργασίας για την ε, πιλωτική λεγόμενη φάση των ομολόγων έργου που στόχο έχει την δοκιμασία, την τροποποίηση και ενδεχομένω την προετοιμασία μιας περαιτέρω πρωτοβουλίας μετά το 2014, στηρίζεται, όπως γνωρίζετε, σε ένα πολύ περιορισμένο ποσό, 230 εκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί για τα ομόλογα έργου, αποτελούν όμως ένα πολύ σημαντικό ε, μέσο μόχλευσης που μπορούν, μπορεί να κινητοποιήσει μέχρι και 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ε, επενδύσεις για τις υποδομές. Το κλειδί για αυτή τη μόχλευση είναι ο καταμερισμός του κινδύνου, πάνω στον οποίο έχουν συμφωνήσει η Επιτροπή με την ε, Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα μοντέλο βάσει του οποίου τα 230 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν ένα πρώτο μέσο ανάληψης κινδύνου μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο ε, επιλέξιμων έργων που υποβάλλεται στην τράπεζα, από την τράπεζα. Και έτσι οι ενδογενείς ελλείψεις στην ε, ε, υποβολή στις προτάσεις αυτές μέσω του χαρτοφυλακίου και η κάλυψη του πρώτου αυτού βήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα 230 εκατομμύρια έχει σαν αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται το ε, ποσό αυτό σαν εγγύηση. Ως εξή. Η τράπεζα θα εκδώσει μια εγγυητική ενίσχυση, ένα δευτερογενές ε, χρέος ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα επιλέξιμα έργα. Με ένα επιπλέον ποσό δευτερογενούς χρέους πάνω από την χρηματοδότηση που προβλέπεται στα έργα, που ε, ως εκ τούτου θα αποτελέσει ένα επιπλέον στρώμα προστασίας. Αυτό το επιπλέον στρώμα προστασίας σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του έργου, που είναι οι δανειζόμενοι στις δομές αυτές, θα μπορέσουν να εκδώσουν ασφαλή ομόλογα με επίπεδο και απόδοση κινδύνου αρκετά ισορροπημένη και ως εκ τούτου ε, ελκυστικά για την κεφαλουργική αγορά. Για την πιλωτική αυτή φάση τώρα. Έχουμε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2012 με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας και προβλέπουμε για την πιλωτική αυτή φάση να στηρίξουμε περί τα 5 με 10 έργα και λόγω βέβαια των χρονικών περιορισμών θα πρέπει να περιοριστούμε, να εστιαστούμε πολύ αυστηρά σε αυτά τα έργα. Δεν έχουμε περιθώριο δηλαδή για υποβολή προτάσεων επιπλέον. Τα έργα με τα οποία έχουμε την ίδια επικοινωνία ενδεικτικά σας αναφέρω. Είναι έργα στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένεται να συναυθεί η πρώτη συμφωνία στο τρίτο τρίμηνο ακόμη και γενικά βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές προτάσεις για έργα. Κάθε τρίμηνο βλέπουμε και νέες προτάσεις. Πρώτα διδάγματα από την πρωτοβουλία και υπογραμμίζω πρόκειται για μια πολύ αρχική φάση. Πάντως πρέπει να πω ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερη αισιοδοξία από την ανταπόκριση και των ε, οργανισμών ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τα ομόλογα. Οι, Moody's, η S&P και η Fitch έχουν ε, και οι, τρεις κύριες, και οι τρεις κύριοι οργανισμοί έχουν δώσει θετική αξιολόγηση. Άρα αυτό είναι λόγος αισιοδοξία, αλλά και από τις αρχές χορήγησης, τους χορηγούς και τους επενδυτές έχουμε θετική ανταπόκριση. Επίσης, άλλα διδάγματα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές, σε παραδείγματι στις ε, ε, εντολής, στις αρχές εντολής, αλλά και σε άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες. Οι αρχές εντολής και οι χορηγοί πάντως αναγνωρίζουν ελκυστικότητα στο έργο τέτοια που είναι διτεθειμένοι να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές. Οι αρχές ανάθεσης αλλά και η χορηγή ως ε, προς τα ποσά και τα χρονοδιαγράμματα. Η πιλωτική φάση λοιπόν όπως είπα είναι εν εξελίξη. Μέχρι τώρα δείχνει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον η αγορά. Δοκιμάστε τώρα το τεχνικό κομμάτι με πραγματικά προγράμματα, με πραγματικά έργα σε τρει-τέσσερι τομεί. Η ανταπόκριση αγορά ήταν πολύ θετική και ιδίω βλέπουμε πολύ καλή ανταπόκριση πλευρά των οργανισμών αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα τέτοια που μας ε, που μας δίνει λόγους να αισιοδοξούμε ότι είναι δυνατόν να λειτουργήσει ικανοποιητικά, αλλά βέβαια περιμένουμε και το πρώτο κύριο ορόσημο, ορόσημο που θα είναι η υπογραφή του πρώτου έργου, της πρώτης συμφωνίας για έργο προς τα το τέλη του δεύτερου τριμήνου του έτους, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό εργαλείο για τη λειτουργία των έργων μέσα σε μια κεφαλουργική αγορά και επενδύσεις που θα επιτρέψουν μια απρόσκοπτη μετάβαση σε ένα ε, ευρύτερο πλαίσιο για τα ομόλογα έργων. Και θα δώσω το λόγο και στο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Θέλω να εστιάσω την προσοχή στα θέματα συμφωνίας συνεργασίας που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εφαρμογή αυτών των μέσων και την, και τη λειτουργία αυτών των μέτρων. Η Συμφωνία Συνεργασίας βασίζεται και αντλεί από μια ολόκληρη σειρά νομικών εγγράφων. Έχουμε την νομική βάση την ίδια, έχουμε τον νέο ε, δημοσιονομικό κανονισμό που κανονικά ισχύει στα δημοσιονομικά μέσα από την 1η Πρώτου 2014. Εμείς έχουμε όμως εξασφαλίσει πως η Συμφωνία Συνεργασίας που υπογράψαμε με την, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τον περασμένο Νοέμβριο ήδη συμμορφούνται προς, ε, τα άρθρα του νέου κανονισμού Προβλέψαμε δηλαδή αυτή την, ε, την ισχύ και τέλος έχουμε και τις νομοθεσίες που, είναι τα επιλέξιμα, που αφορούν τα επιλέξιμα προγράμματα που μπορούν να, να ωφεληθούν από τις πρωτοβουλίε αυτές. Έχουμε δουλέψει λοιπόν με δραστήριο τρόπο ώστε να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία συνεργασίας ε, με όλα τα στοιχεία τα οποία ε, περιλαμβάνονται στον ε, ε, δημοσιονομικό κανονισμό προς χάρη του χρόνου ε, οικονομίας Χρόνου. Ο Νίκα εξήγησε ήδη τους στόχους γιατί τους γνωρίζετε, γιατί το Κοινοβούλιο είναι ένας από τους υποστηρικτές της ε, πρωτοβουλίας για τα ομόλογα έργου και όσον αφορά τη διαχείριση του προπολογισμού πιστεύω πως για τα πιλωτικά προγράμματα χρειάστηκε να εξασφαλίσουμε δύο διαδικασίες. Όπως γνωρίζετε έχουμε οικονομικούς πόρους που προέρχονται από τα ο προπολογισμό τι και τεν e. Μετά έχουμε τα δίκτυα για την ενέργεια και για την ε, πληροφορική τεχνολογία και έχουμε μια πίστοση υποχρεώσεων για το 2010 αλλά για την συμβολή ε, ε, των δικτύων τι για να μην μείνουν να χρησιμοποιεί τη δημοσιονομική πόρη. Έχουμε κάνει μόνο μία υποχρέωση, μια αρχική μικρή πληρωμή και μετά θα καταναμηθούν αυτά όταν και εφόσον ε, ε, χρειαστεί δέσμευση των πόρων και υπάρξουν υπογραφές. Αποφύγαμε δηλαδή για το TEN TAF να έχουμε στην σειρά οικονομικούς πόρους οι οποίοι κάθονται σε λογαριασμούς. Χρειάστηκε να ε, κρατήσουμε ξεχωριστούς υποπροϋπολογισμούς έτσι ώστε η Δημοσιονομική Αρχή να γνωρίζει ακριβώ του πόρου που χρησιμοποιούνται για τι μεταφορέ, αυτού που χρησιμοποιούνται για την ενέργεια κτλ. Ε, η εφαρμογή έτσι γίνεται πιο περίπλοκη κάπω, αλλά είναι σύμμορφη προ την, ε, την ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Έχουμε χωριστέ γραμμέ του προπολογισμού και γι' αυτό η κάλυψη των απολειών των ζημιών σαφώ θα αποδοθεί στι ζημιέ, αν αυτό χρειαστεί δεύτερον και επόμενο σημείο είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια ειδική διαδικασία για την επικύρωση της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων. Και νομίζω πως ε, όταν θα έχει θεσπιστεί πλέον η επιλεξιμότητα, η τράπεζα είναι υπεύθυνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε ε, πρόγραμμα. Για κάθε τομέα λοιπόν υπάρχουν ε, συγκεκριμένα δελτία επιλεξιμότητας ε, της πολιτικής που εγκρίνονται από την Κομισιόν έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε στήριξη από αυτά τα προγράμματα και από αυτή την πρωτοβουλία θα συμμορφώνεται προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά ορίζονται από την Κομισιόν σε συνεργασία με τις πολιτικές ε, αρχές για την ε, κοινή ανάληψη κινδύνου ε, καλύπτουμε, το κίνδυνο από πλευρά τη Κομισιόν να έχουμε ευθυγράμμιση συμφερόντων και να είμαστε βέβαιοι πω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προβαίνει στη σωστή εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου που μπλέκεται και γι' αυτό καλύπτουμε μόνο το 95% και ενώ η τράπεζα καλύπτει το 5% για να είμαστε βέβαιοι ότι θα φροντίσει τους πόρους μας όπως φροντίζει τους δικούς της πόρους. Και επιπλέον φυσικά στο ισοζύγιο τους, στον ισολογισμό τους μάλλον, ε, ε, ε, αναλαμβάνουν και τον υπολοιπόμενο κίνδυνο. Αυτά είναι μέσα στις αρχές της, του, της υγιούς νοσονομικής διαχείρισης όπως θεσπίζεται από τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό για τα νέα δημοσιονομικά μέσα μετά το 2014. Υπάρχουν βέβαια διάφορες... Άλλες συμβατικές ρήτρες για την διακυβέρνηση Και νομίζω για τη διακυβέρνηση η Διευθύνουσα Επιτροπή που εμπλέκει και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δώσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να έχουμε διορθωτικές δράσεις εάν υπάρξει ανεπαρκής απόδοση, αν υπάρχουν άλλα προβλήματα προς επίλυση. Λοιπόν, η διακυβέρνηση αυτή προβλέπει ένα μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης για τις αμοιβέ και της, ε, ε, των εμπλεκομένων. Έχουμε ένα διοικητικό τέλος που καλύπτει το βασικό κόστος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα σχέδια αυτά, αλλά υπάρχει και πρόσθετη επιβράδυνση, ένα πριμ απόδοσης που θα δώσει κίνητρα στην Τράπεζα Επενδύσεων να λειτουργήσει σε περισσότερες χώρες. Αντί να έχουμε λοιπόν ένα ποσό κατά που δεν δίνει καμία έμφαση στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να έχει σχέδια σε πολλούς τομείς και σε πολλές χώρες. Έχουμε μια δομή ανταμοιβών που οδηγεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο να προτάξει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την χρήση ως το δυνατόν περισσότερο των κονδυλίων σε διάφορους τομείς και φυσικά και με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό έχουμε συμπεριλάβει όλες τις πρόνοιες σε σχέση με την ορατότητα και τη διαφάνεια που είναι απαραίτητες μέσα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης τις ρήτρες του δημοσιονομικού κανονισμού για την σωστή και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κτλ. και έχουμε και μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε έξι μήνες. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα πιλωτικό σχέδιο λοιπόν, προσπαθούμε να είμαστε προορατικοί και εξασφαλίσουμε τα καλύτερα πιθανά πρότυπα. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν έχουμε ενώπιόν μας την πραγματική δοκιμασία να υπάρξουν πραγματικά έργα τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε όσο το περισσότερο περισσότερα τέτοια σχέδια εν ώψη της δύσκολης μακροοικονομικής συγκυρίας για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια γιατί η καθυστέρηση, η επιβράδυνση των ε, ε, δημοσίων επενδύσεων, όπως είπε ο κ. Τσέινεμ, έχει δημιουργήσει και προβλήματα στις ιδιωτικές επενδύσεις και έχουμε προσπαθήσει μαζί με την, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχουμε κοινέ ενέργειες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα καθυστερήσεων σε διάφορα σχέδια και έτσι θα μπορέσει να μας βοηθήσει να υπερκεράσουμε τις αμφιβολίες κάποιων επενδυτών και να έχουμε επιτυχή προγράμματα. Ο ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά και Γενικέ Διευθυντά για τις σαφείς παρατηρήσεις σας και παρουσιάσεις. Αν μπορούμε να κάνουμε μία αεροναυτικού χαρακτήρα σύγκριση αυτών των ε, εξελιγμένων προϊόντων, είναι σαν να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχέτυπο και είμαστε στη φάση του roll-out, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Βγαίνει το πιο πρώτο αρχέτυπο από το εργοστάσιο και τώρα πρέπει να πετάξει. Πάντως έχουμε βγει από το επίπεδο σχεδίασης, επί χάρτου εργάζεται το αεροπλάνο, αλλά πρέπει να πετάξει. Ο Γκέραν Φέρμ, ο οποίος είναι ο ειδικός για τα μηχανολογικά, Ευχαριστώ. Δεν είμαι μηχανικό. εν πάση περιπτώσει ήμουνα ο εισηγητή για αυτό το θέμα και έκανα τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για να ξεκινήσουμε σε αυτή την πιλωτική φάση. Μετά από αυτά που ακούσαμε, έχουμε μια επιβεβαίωση για αυτά που είπαμε στην εκθεσή μα, ότι αυτό είναι πράγματι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία λαμβάνει, κάνει τα απαραίτητα για να γεμίσει ένα κενό στην αγορά, που θα είναι πολύ σημαντικό από ό,τι βλέπω από τι τεχνικές πτυχές τη Συμφωνία Συνεργασία συνάδει και με τις προϋποθέσεις που θέσαμε και στη δική μας έκθεση για τα θέματα αυτά. Και το ίδιο ισχύει για το γεγονός ότι είναι απόλυτα α, συνάδων και με το δημοσιονομικό κανονισμό. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό θέμα είναι η επιλογή των σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν και αυτό πρέπει να το κάνουμε με σωστό τρόπο για να εξασφαλίσουμε και την ε, να καταδείξουμε και τη σημασία του εγχειρήματο. Από ό,τι ξέρω από τις χρηματαγορές και τους επενδυτές, επενδυτές, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά σχέδια υποψήφια, αλλά θα πρέπει να επιλέξουμε αυτά τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την αγορά. Τα οποία είναι κοντά στην ικανότητα χρηματοδότηση από την αγορά, αλλά όχι αρκετά καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι βιώσιμα αυτά τα σχέδια. Κατανοώ ότι πρέπει να έχουν φτάσει σε ένα αρκετά προχωρημένο ε, επίπεδο, γιατί είναι περιορισμένο το χρονικό όριο που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι κίνδυνος όμως ότι θα είναι δύσκολο να καταδείξει κανείς πόσο σημαντικά είναι αυτά τα σχέδια. Αν είναι πολύ καλά, αν είναι πάρα πολύ καλά, θα έπρεπε να τα έχει χρηματοδοτήσει η αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τα σχόλια σας για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε βιώσιμα σχέδια. Αν δεν μπορούμε όμως να αποδείξουμε ότι βρήκαμε κάποια σχέδια που η αγορά δεν θα τα χρηματοδοτούσε και ήταν κεφαλαιόδης η δική μας συνεισφορά, θα είναι πολύ σημαντικό να τα αποδείξουμε. Δεύτερο ερώτημα για τις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση των υποδομών έχει περικοπεί σημαντικά, το Connecting Europe έχει μειωθεί, στα μισά περίπου και λιγότερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τομέα της ε, ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνολογίας πληροφοριών. Εκεί θέλει να κόψει το Συμβούλιο και να πετσοκόψει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέμε να τους αποδείξουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμα σκεπτικισμός σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά είναι απαραίτητο να αποδείξουμε στο Συμβούλιο ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικά. Αυτά που λένε ορισμένε φορεί πιστοληπτική αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικά. Αλλά τι γίνεται τώρα για να αντιμετωπίσουμε το σκεπτικισμό που υπάρχει στο μυαλό ορισμένων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στο Συμβούλιο για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι όλα αυτά είναι απολύτως σημαντικά και απαραίτητα. Και έρχομαι στο τρίτο μου σημείο στην παρουσίαση της Κομισιόν για τη διαχείριση του προϋπολογισμού είπε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες, μία για τα TNT και η άλλη για την ενέργεια και τις τεχνολογίες πληροφορίας. Στο δεύτερο τμήμα υπάρχει μόνο ένα σχέδιο που μπορεί να χρηματοδοθεί ή ενέργεια ή τεχνολογίες πληροφοριών. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι η πιλωτική φάση θα δουλέψει και στους τρεις τομείς και μεταφορές και ενέργεια και τεχνολογίες της πληροφορίας. Αν έχουμε μόνο ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο στους τελευταίους δύο τομείς, πώς θα αποδείξουμε αυτή την βιωσιμότητα και στις δύο αυτές περιοχές. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, θα πρέπει να έχουμε σε όλους τους τομείς σχέδια για να αποδείξουμε και τη σημασία της πιλωτικής φάσης σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτές είναι λοιπόν οι αντιδράσεις μου σε αυθόρμητο επίπεδο για τις πιο τεχνικές λύσεις. Δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα θέματα, η επιλογή των σχεδίων και ιδίως η κάλυψη και των τριών τομέων και η διακρύβωση και απόδειξη της σημασίας της πιλωτικής φράσης, όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Σας. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Το ερώτημα και τα επιχειρήματα που Νομίζω ότι είναι προς προς τα όσα είπε ο κύριος Φέρν. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα ομόλογα έργου να καλύψουν ε, την ανάγκη για ένα καινούριο μέσο, ένα μέσο το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει αγορά. Και ίσως να μην έπρεπε να το πω αυτό που θα πω, αλλά συνήθως ε, σας ασκούνται πολλές πιέσεις να προχωρείτε γρήγορα και αν τελειώνετε εγκαίρως ε, το έργο που σας αντιστοιχεί και γενικώ το πρόβλημα είναι ο χρόνος. Για μένα ως πολιτικό όμως είναι πολύ σημαντικό τώρα αντί για το χρόνο να κάνουμε τη δουλειά πολύ σωστά. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτό το κύριο μήνυμα που θέλω να σας απευθύνω και τι μπορεί να συνεπάγεται και κάποιες καθυστερήσεις. Πάντως με εντυπωσίασε το ότι αναφέρατε κάποια έργα που βρίσκονται σε πιλωτική φάση Ε, μπαίνω με κατηγορούν πάντα στην πατρίδα μου ότι θέλω να στρώλω τα πάντα με άσφαλτο. Μ' αρέσουν πολύ αυτοκινητόδρομοι. Ναι, ναι, μ' αρέσουν και θέλω να έχω κι άλλους. Αλλά βλέποντα εδώ στον κατάλογό σας μου κάνει εντύπωση ότι μόνο για αυτοκινητοδρόμου μιλάτε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν επενδύσεις ε, σε ράγα, σε σιδηρόδρομο. Εκεί που είναι πιο δύσκολο δηλαδή να βρεθεί η χρηματοδότηση από την αγορά. Ή στην ενέργεια στις ανεμογεννήτριας. Άρα δεν θα, πρέπει να, δεν θα πρέπει εσείς να επιλέξετε εκείνα τα έργα τα οποία είναι πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθούν από την αγορά. χρηματοδότηση των αυτοκινητοδρόμων τη βλέπουμε να γίνεται από την αγορά σχετικά εύκολα στα κράτη-μέλη. Αυτό το μήνυμα λοιπόν θα σας απέστειλε εγώ. Είναι πολύ σημαντικό το νέο μέσο που θα οικοδομήσουμε να προσφέρει προϊόν το οποίο δεν προσφέρει αγορά. Και επαναλαμβάνω να δώσετε αρκετό χρόνο στον εαυτό σας ώστε να το προετοιμάσετε σωστά. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ο κύριο Ρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν, αλλά τα υποστηρίζω πλήρω τα λόγια. Και αν και του Γκέραν. Για το πόσο μεγάλη σημασία έχει και η ποιότητα εδώ. Μια ερώτηση, τόσο προς εμάς και προς την Επιτροπή. Αν έχουμε να κάνουμε ένα πιλωτικό έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε τέλη του 2014 και που θα πρέπει να υποβληθεί σε μια αξιολόγηση. Γιατί κάποια στιγμή σταματάνε τα πιλωτικά έργα, έτσι γίνεται η διακοπή ενδεχομένως εκτέλεση. Ε, και πρέπει θεωρητικά μέσα σε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και με νέε διατάξει ενδεχομένω να γίνει η αξιολόγησή του. Ε, αυτό λοιπόν θέλω να μάθω. Τι θα συμβεί με τα πιλωτικά προγράμματα μέσα στην ε, χρονική προθεσμία που προβλέπεται για την αξιολόγηση θα μπορέσουν η Επιτροπή και η ΕΤΕ να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση. Σε ποια χρονική στιγμή θα γίνει αυτή, με ποια διαδικασία θα επανέλθουν ανάπιον Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ώστε να ζητήσουν την επικύρωση αυτού του πιλωτικού έργου, ώστε να γίνει ένα μόνιμο μέσον. Και μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη ακόμη είναι πολύ επιφυλακτικά απέναντι σε αυτό. Μεγάλα λοιπόν τώρα ατοματικά, δεδομένου ότι αυτό θα συμβεί κάπου στις, στα τέλη του 2014 αυτή η αξιολόγηση. Ερωτώ λοιπόν τι συμπεράσματα, πότε θα έρθουν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, τι θα προτείνει η αξιολόγηση με βάση τα, τα συμπεράσματα και τι θα γίνει δεδομένου ότι μπορεί να μην υπάρχει το σχετικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε να, να τροφοδοτούμε το σύστημα με έργα, θα τα προβάλλουμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να ε, θέσει τα ερωτήματά της Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα έργα και πάλι. Και δεύτερη ερώτηση. Η μόχλευση. Υπάρχουν δύο ορόσημα στο φαινόμενο της μόχλευσης που να μας επιτρέπουν να πούμε ότι κάτω από αυτό και πάνω από εκείνο το ορόσημο δεν έχει λόγο ύπαρξη στο ομόλογο έργο. Εάν ας πούμε είναι υπερβολικά υψηλή η μόχλευση, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, μήπως σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο και μήπως τότε ένα τέτοιο δημοσιονομικό μέσο δεν είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί και είναι σκόπιμο τώρα κάποιο άλλο. Ή εάν είναι επί 40 η μόχλευση, μήπως τελικά δεν αρκεί μόνη της η αγορά. Άρα, ναι, μήπως θα έπρεπε η αξιολόγηση να ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση, αλλά από την άλλη πως πρέπει και η Επιτροπή και η ΕΤΕ να ορίσουν αυτό και το όριο. Ανάλογα με τις δυνατότητες, με την επάρκεια της αργοράς ή του έργου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ζητάει το λόγο. Α, μάλιστα, ο κύριος Φάρμ. Ξέχασα κάτι. Υπάρχει μια συγκέντρωση στο κατάλογο που μας είπατε για τους αυτοκινητόδρομους. Μια άλλη γη. Υπάρχει και μια γεωγραφική συγκέντρωση στα πλουσιότερα κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Βέλιο. Αυτό μας ανησυχεί. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι βιώσιμη αυτή η πρωτοβουλία, όχι μόνο στα πλούσια κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Τι κάνετε για γεωγραφική ισορροπία, υπάρχει κάτι το οποίο έχετε προβλέψει. Δεν υπάρχει κανένα άλλο τώρα πια. Μπορούμε να ξαναδώσουμε το λόγο στην Κομισιόν και στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να απαντήσουν το ερώτημα και να εξηγήσουν γιατί πονάχα ένα ενεργειακό πρόγραμμα ή τηλεπικοινωνιών και γιατί εστιάζουμε στους αυτοκινητοδρόμους και επιπλέον στις πλούσιες και δυτικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τι γίνεται μετά την πιλωτική φάση και ποια είναι η προβλεπόμενη μόχλευση. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Από την πλευρά της Κομισιόν. Ξεκινώ από το τέλος. Και θα γυρίσω ανάποδα. Τι θα γίνει μετά την πιλωτική φάση. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ως τμήμα της, ε, έχουμε δεσμευτεί να υπάρχει μια ενδιάμεση αξιολόγηση στο τέλος του 2013 και μετά μια συνολική αξιολόγηση που θα γίνει στο τέλος του 2014. Θα υποβάλουμε λοιπόν αυτές τις εκθέσεις και θα έχουμε και μια εξωτερική αξιολόγηση για την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Η θέση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με την πρωτοβουλία αυτή στη νέα περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Προβλέπουμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία από το 2014 και η τελική αξιολόγηση που θα έρθει στο τέλος του 2014 θα πρέπει να προσαρμόσει τις δεσμεύσεις οι οποίες τις δεσμεύσεις οι υποχρεώσεων που θα γίνουν είτε συνολικά είτε κατά τομής για τη συνέχεια, αλλά βάσει τις αναλύσεις που κάνουμε στην αρχή της διαδικασίας και με την ενθάρρυνση της αγοράς θα ήταν πιστεύουμε αντιπαραγωγικό να κάνουμε αυτό που είπε ο αξιότιμος κύριος Βουλευτής, να στα... κάνουμε αυτό το πρόγραμμα για ένα χρόνο, μετά να σταματήσουμε και μετά να ξαναρχίσουμε, να προσπαθήσουμε να ξαναρχίσουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτά που λέτε και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, έρχομαι σε ένα από τα πρώτα σχόλια που έγιναν για την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν σχέδια που η αγορά δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει αλλά έχουν προσθέμενη αξία η έννοια της προσθέμενης αξίας είναι πολύ σημαντική για την Κομισιόν και θα επιμείνουμε πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Αλλά είναι μια προσθέμενη αξία διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούμε στα πιο μεγάλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε από την άποψη ότι έχουμε έργα τα οποία χρειάζονται χρηματοδότηση. Με τις αναλύσεις μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς δανειοδότησης ή δανειοδότησης με άλλους τρόπους για τα σχέδια αυτά. Η λογική μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι με τη δική μας παρέμβαση μπορούμε να προσελκύσουμε επενδυτές κεφαλαιοαγορές, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες να χρηματοδοτήσουν αυτά τα σχέδια και επομένως να προσελκύσουμε επενδυτές οι οποίοι αλλιώς δεν θα ενδιαφερόταν. Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση στην οποία θα πρέπει να προβούμε γιατί προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία των project bonds για να έχουμε νέες μορφές επενδυτών στις ευρωπαϊκές υποδομές, αλλά δεν χρηματοδοτούμε εμείς αυτά τα σχέδια υποδομών. Αναζητούμε τους ε, ιδιώτες επενδυτές και γι' αυτό περιοριζόμαστε σε αυτά τα οποία δεν κάνουν ήδη μόνοι τους. Εμείς επεμβαίνουμε για να επιτρέψουμε να έρθουν άλλοι ιδιωτικοί πόροι που δεν είναι τραπεζικού χαρακτήρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο στόχος μας είναι να πείσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Και είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό αν τους πούμε ότι έχουμε πολλά σχέδια για φέτος, αλλά για δύο χρόνια δεν έχει τίποτα. Και μετά έχει ο Θεός, μετά το 2016. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η συνέχεια γιατί η ασυνέχεια θα αποτρέψει τους επενδυτές οι οποίοι μέχρι τώρα δεν επένδυαν σε ευρωπαϊκά σχέδια υποδομών και τώρα περιμένουμε από αυτούς να έρθουν να καλύψουν αυτό το χώρο. Από την πλευρά της Κομισιόν θεωρούμε λοιπόν ότι η συνέχεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το τελικό θέμα για την κατατομή και τη γεωγραφική κατανομή. Πιστεύουμε στην Κομισιόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερα φάσματα σε γεωγραφικό και τομεακό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο έχουμε γι' αυτό έχουμε δώσει ισχυρά κίνητρα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορους τομείς και να έχουμε μια ευρύτερη γεωγραφική κατανομή γιατί αλλιώ δεν θα υπήρχε αυτή η κάλυψη του απαραίτητου κόστου. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ισχυρά κίνητρα. Από την άλλη πλευρά είναι και πάλι σημαντικό να ξέρουμε ότι εφέτος θα τρέξει το πιλωτικό σχέδιο και τα σχέδια τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι σχέδια τα οποία πρέπει να έχουν ήδη ξεκινήσει στο παρελθόν γιατί είχαν γίνει οι μελέτες σκοπιμότητος, μελέτες επίπτωσης στο περιβάλλον και ξέρετε επομένω ότι τα σχέδια αυτά υποδομών δεν ξεκινάνε σε ένα μήνα και σε έξι μήνες να είναι έτοιμα για χρηματοδότηση. Επομένως, για τα πιλωτικά σχέδια, το χρονικό διάστημα προετοιμασίας καθορίζεται από τις δημόσιες αρχές της κάθε χώρας και καθορίζεται και από το γενικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μέσα σε αυτά τα όρια κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να παροτρύνουμε και να οθήσουμε τους επενδυτές να έχουν κίνητρα να κάνουν πράγματα. Και εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και εγώ νιώθω ιδιαίτερα ενθαρρυμένος αλλά και σπρωγμένος από την Κομισιό. Συμφωνούμε στο σημείο αυτό. Το μόνο που θέλω να προσθέσω, αυτά που είπε ο κύριος Τόμας, είναι ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το καινοτόμο του εγχειρήματο. Προσπαθούμε να επιτύχουμε κάτι το οποίο είναι μια σημαντική συνεισφορά σε μια δημιουργία μιας νέας μορφής ενεργητικών στην Ευρώπη. Μέσω της αγοράς και όχι κόντρα στην αγορά. Αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα. Πρώτα, ότι αυτό το εργαλείο κινείται από τη ζήτηση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να απαντήσει μόνο στι προτάσει που θα τι υποβληθούν, μόνο στι προτάσει που θα προέλθουν από την, το ιδιωτικό τομέα και θα έχουμε κάποιε ενδείξει θετικέ από του φορεί πιστοληπτική ε, αξιολόγηση και από την αγορά. Όλα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα για να μα βοηθήσουν να επιλέξουμε. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι η πιλωτική αυτή φάση εξασφαλίζει ότι έχουμε θεσμούς που είναι επιφυλακτικοί σε σχέση με την ε, είσοδο σε αυτό το νέο τομέα χρηματοδότησης ενεργητικών. Επομένως, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να ξεκινήσουμε ώστε να δούμε περισσότερα πιλωτικά προγράμματα για να καταδείξουμε ότι η τεχνολογία αυτή λειτουργεί, ότι η οικονομική λογική λειτουργεί, ότι λειτουργούν όλα σε νομικό επίπεδο και είμαι πεπισμένος ότι αν μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά στην πιλωτική φάση, τότε στην γενικότερη προσφυγή στα θέματα αυτά θα έχουμε εξασφαλίσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ όλων των θεσμών για περισσότερα σχέδια. Και αν μου επιτρέπετε ένα ακόμα πράγμα να πω και να ξαναπώ ότι η σημασία αυτού που είπε ο κ. Στομάς είναι πολύ σημαντική. Επειδή προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε χορηγού στο δημόσιο τομέα, και τα διάφορα τους διάφορους θεσμικούς επενδυτές, τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία είναι κεφαλαιόδης να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε μια συνέχεια ή τουλάχιστον την, ευκαι... την προοπτική μιας συνέχειας. Δεν μπορούμε να τους πούμε περιμένετε 18 μήνες ώσπου να αποφασίσουμε. Δεν λειτουργεί έτσι η αγορά οι ομάδες που έχουν αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείε και τα συνταξιοδοτικά ταμεία που είναι οι εταίροι μας δεν θα περιμένουν. Θα πάρει κάπου αλλού. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ λέει η πρόεδρος. Όλα αυτά είναι εξόχως ενδιαφέροντα σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες να ανταγωνιστούμε τις ε, αγορές και εάν θέλουμε πραγματικά να πείσουμε τις, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συνταξιοδοτικά ταμεία να επενδύσουν εκεί και όχι στην αγορά, δεν ε, θα είναι εύκολο αυτό αν δεν έχουν και τα, την απαραίτητη απόδοση. Από την άλλη πλευρά, τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουμε ενώπιόν μας είναι μακρόπνοα πρόγραμματα. Και ας σκεφτούμε πόσο κρατάνε οι κατασκευές αυτοκινητοδρόμων, χρειάζονται πολλές διαδικασίες αξιολόγησης, ε, δοκιμασιών κτλ. Όλα αυτά είναι σαφή. Εν πάση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι παροτριμένη μεν, αλλά σπρωγμένη δε. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε ότι μαζί με την Κομισιόν θα προχωρήσετε όλα αυτά τα σχέδια. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό ταξίδι. Επιστροφής. Επόμενο σημείο. Πρέπει να σκεφτούμε και για την εντολή μας και την ομάδα διαπραγματεύσεων για το προϋπολογισμό του 2014. θα, θα ζητήσω τώρα από την Αν να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ψηφίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την δημοσιονομική διαδικασία την περασμένη εβδομάδα. Και όπως θα θυμάστε, θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Και επίσης, όπως θυμάστε, ψηφίσαμε διάφορα σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα προκύψουν στο τριμερή διαλόγο με το Συμβούλιο. Καταρχήν τη σχέση ανάμεσα στον προπολογισμό του 2014 με το πολιετές νομοσυνομικό πλαίσιο το οποίο ήδη ανέφερε ο κύριος Ρικέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε τι θα χρησιμοποιήσει ως βάση η Κομισιόν για να προτείνει τον προϋπολογισμό του 2014. Αυτό αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης. Υπάρχει ολόκληρη υπόθεση των πληρωμών και των προβλημάτων που έχουμε με τα ρέστα και τα προβλήματα που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια πληρωμών που μετακυλίονται από τη μια χρονιά στην άλλη και φοβόμεθα πως θα υπάρξει μια χιονοστιβάδα με πληρωμένων υποχρεώσεων που θα, ανα... που θα μας έρθουν και θα μας κατακλείσουν και πριν αρχίσει το 2014 ε, δηλαδή θα έχουμε ένα σωρό πληρωμές από το 2013 και έπειτα ζητάμε ε, από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να φτιάξουν μια ομάδα εργασίας που θα εξετάσει τις ε, εξελίξεις σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε να έχουμε μια καλύτερη διαδικασία από ό,τι σε άλλα χρόνια, να αρχίσουμε δηλαδή να χειριζόμαστε το θέμα με πιο ρεαλιστικό τρόπο και έχουμε και τις πολιτικές μας προτεραιότητες που φυσικά συνδέονται με τη στρατηγική 2020. Επίσης το Συμβούλιο πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές που κάνουν λόγο για ανάπτυξη, για περικοπές ε, και θα έχουμε ένα τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό που προβλέπεται για τις 19 Μαρτίου. Και πέρα από τα όσα αναφέρονται εδώ, στις κατευθύντριες μας γραμμές σε σχέση με την εργασία για τις πληρωμές και τα ραλ, θα είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση για το πώς και τι θα κάνουμε με την ετήσια δημοσιονομική διαδικασία, όπως το έχουμε συζητήσει και παλιότερα, τι είδαμε τις περασμένες φορές, μάλλον τα όσα είδαμε τις περασμένες φορές δεν ήταν πολύ ωραία, όλα φαίνεται να γίνονται τελευταία στιγμή, μετά από τη δική μας ψηφοφορία, ε, ετοιμάζεται το Συμβούλιο για Διαπραγματεύσεις. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα τα καταφέρουμε ώστε να γίνει σωστή συζήτηση και ίσως και πιο λεπτομερή συζήτηση νωρίτερα. Αυτά νομίζω θα πρέπει να κάνουμε για τον τριμερή διάλογο. Αυτές οι κατευθυντήρες στις οποίες συμφωνήσαμε θα πάνε στην Ολομέλη, θα τις ψηφίσουμε και μετά η διαδικασία είναι ότι θα γίνει ο τριμερής διάλογος περί προπολογισμού στις 19 Μαρτίου και στη συνέχεια η Κομισιόν θα παρουσιάσει το σχέδιο προπολογισμού στα τέλη Απριλίου. Ανακοίνωσαν πως θα το υποβάλλουν ε, σε κάποια εβδομάδα που δεν θα έχουμε συνεδριάσει στο Κοινοβούλιο. Πράγμα που είναι κάπως παράξενο, διότι συνήθως έχουμε μια παράδοση ότι η Κομισιόν έρχεται και παρουσιάζει τον προπολογισμό στο Κοινοβούλιο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να θέτουμε ερωτήσεις και νομίζω πως η Κομισιόν θα πρέπει να αναθεωρήσει τα σχέδιά της και να βρει κάποια άλλη ημερομηνία ώστε όταν δηλαδή το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας συνεδριάζει. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή έχει, νομίζω, ήδη ξανασυζητήσει, ξανασκεφτεί καλύτερα την ημερομηνία. Το ανέφερε και ο Άλλα. Ήδη διατυπώνονται κάποιες αμφιβολίες. και ε, με τη βάση ότι το, για το 2014 ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλυθεί σε κάθε χωριστή γραμμή για να συζητηθεί. Άλλος Αιντα. Όπω έλεγε η Αίντα. Όπως έλεγε η κυρία Γένσεν, αυτό που εγκρίναμε ήδη στην Επιτροπή μας και φυσικά θα εγκριθεί και στην Ολομέλεια, θα καθορίσει τις προτεραιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να ξεκινήσει την επεξεργασία του προϋπολογισμού. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα ποια ακριβώς θα είναι η πρόταση της για τον προϋπολογισμό, σε ποια αριθμητικά στοιχεία θα βασίζονται. Αυτό το οποίο δεν είναι άγνωστο είναι τα προβλήματα των πληρωμών που ήδη τα σέρνουμε από τα προηγούμενα χρόνια και θα τα αντιμετωπίσουμε και εφέτος. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό των 16 ε, δισεκατομμυρίων που έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια και το κόστος επίσης των, ε, του κενού που θα δημιουργηθεί το 2013 και θα μεταφερθεί στο 2014 και στο δημοσιονομικό πλαίσιο των επομένων έτων. Αλλά γενικά οι πολιτικές ομάδες έχουμε συμφωνήσει για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τη συναντρίαση του Μαρτίου και θα δούμε στη συνέχεια. Ντομινίκ. Ένα ερώτημα μονάχα. Τη στιγμή που δεν ξέρουμε ούτε πώς ούτε πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014, σε τι συνίσταται το νόημα της συνεδρίασης του τριγωνικού διαλόγου. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα συζητήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Ε, εφόσον δεν θα έχουμε ουσιαστικά πρόταση της Κομισιόν. Πάντα είναι έτσι στις διαδικασίες προϋπολογισμού. Ο πρώτος τριγωρικός διάλογος με την Προεδρία του Συμβουλίου γίνεται προτού να διατυπωθεί το πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού από το προσχέδιο προϋπολογισμού καλύτερα από την Κομισιόν. Πάντα κάνουμε ένα τρίλογο, τριάλογο αυτού του είδους λένε οι εισηγητές ποια είναι η εντολή τους, ποιες είναι οι κατευθυντήρες γραμμές τους. Το Συμβούλιο λέει ποια είναι η δική του άποψη, λέει ότι κατανοεί αυτά το οποία λένε οι εισηγητές, λέει ότι θα συνεργαστεί μαζί μας και μετά κάνουν του κεφαλιού τους. Ποιος ξέρει όμως, μήπως αλλάξουν φέτος τα πράγματα αυτά. Εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξη, ίσως το Συμβούλιο για μια φορά να καταφέρει να σκεφτεί επί τη βάση αρχών, κατευθυντηρίων, γραμμών, να διατυπώσει ακόμα και τις δικές του προτεραιότητες στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει τα ίδια προβλήματα, ότι και το ίδιο δεν μπορεί να ξέρει πώς θα είναι ο προϋπολογισμός που θα προταθεί από την Κομισιόν. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξέρει. Ο καθένα λέει ότι δεν ξέρει τίποτα. Βέβαια και η Κομισιόν η ίδια η οποία θα πρέπει να υποβάλει τον προπολογισμό και αυτή νύπτη τα σύρα τη λέει δεν ξέρει τίποτα. Θα δούμε όμω. Ο κ. Πρίστη ίσω μπορεί να μα πει κάτι για όλα αυτά τα θέματα, να μα δώσει κάποιε κάποιο γενικό περίγραμμα του χρονοδιαγράμματο για το πότε μπορούμε να προσδοκούμε ένα σχέδιο προπολογισμού, ένα προσχέδιο προπολογισμού από την Κομισιόν. το λέω τώρα. Μεταξύ μας κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω να θίξουμε το θέμα της νομικής βάσης ε, για τον προϋπολογισμό αυτό. Απλώς να βασιστούμε σε αυτή που έχουμε τώρα, γιατί στο τέλος θα αναδυθεί αυτό το θέμα, αλλά το να θέσουμε τώρα θέμα νομικής βάσεως, αυτό θα παρατείνει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία αντιπαράθεσης με το Συμβούλιο που έχουμε ενώπιον μας. Και εσείς φυσικά δεν μπορείτε να έχετε τώρα μια ε, νομική βάση τη στιγμή που δεν ξέρετε τι θα προκύψει τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχολιάκια είναι σωστή η ανάγνωσή σας βέβαια για το ρόλο του πρώτου τριγωνικού διαλόγου πριν παρουσιαστεί το σχέδιο προπολογισμού από την Κομισιόν. Η λογική είναι ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν προηγουμένως εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του 2014 και η Κομισιόν θα πρέπει να τις λάβει υπόψη αυτές τις ε, κατευθύνσεις στην προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμών. Το γεγονό ότι υπάρχει μια προηγούμενη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο σκελών τη αρχή του προπολογισμού μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε κάποια σημεία από τι δύο πλευρέ τη αρχή αυτή είτε όχι. Αυτό δίνει και κάποιε ενδείξει και κάποια κατεύθυνση στην Κομισιόν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι μια σημαντική και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και κατά δεύτερο λόγο είναι σημαντικό να τονίσω ότι αυτό είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαφής και η διαδικασία του ετήσιου προϋπολογισμού που θα ακολουθείτε για το 2014, πώς θα γίνει το χρονοδιάγραμμα για τα βήματα που θα ακολουθήσουν ώστε κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να προετοιμάσει την θέση του και τη διαδικασία και έτσι αποκομίζεται η προβλεψιμότητα για την διαδικασία προϋπολογισμού. Από την πλευρά της Κομισιόν υπάρχουν προβλέψεις των συνθήκων για το χρονοδιάγραμμα. Είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα από τις συνθήκες για την τελική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να παρουσιάσει η Κομισιόν τον προϋπολογισμό. Η Κομισιόν θα σεβαστεί φυσικά αυτό το, αυτή την πρόνοια των συνθήκων. Πέραν αυτού του επίσημου χρονοδιαγράμματος υπάρχει και ένα πραγματιστικό χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει πολύ πιο πρόημα την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Κομισιόν ούτως εχόντων των πραγμάτων σήμερα βέβαια μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση ορισμένων εβδομάδων σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα τη Κομισιόν και η Κομισιόν προσπαθεί να ερμηνεύσει τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει σαφές ότι δεν υπάρχει κοινή θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Επί τη βάση αυτή λοιπόν η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα να προετοιμάσει το σχέδιο προπολογισμού τη με βάση αυτών των ενδείξεων, αλλά η Κομισιόν θα σεβαστεί προφανώ τι προδιαγραφέ των συνδικών και το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, καλά. Τότε, αν έχουμε για 1η Σεπτεμβρίου το σχέδιο προπολογισμού, θα πρέπει και με, τις, ε, με την αυτόματη παράταση των ε, νομικών βάσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα περιμένουμε να δούμε τι εκπλήξεις θα μας ετοιμάσετε. Πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα κάπως ε, ε έδαφος, για να μην πω ασταθές. Εάν δεν υπάρχει όμως άλλος συνάδελφος να στήσει το λόγο, ίσως η συγγήτρια μπορεί να μας πει αν έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις της, τις προσωπικές, για το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης και την πολιτική για τα κτίρια, κυρία Χολμαϊρ. αφού μας απασχόλησε τόση ώρα το πολιτές νομικό πλαίσιο και όλα αυτά τα θέματα, ας περάσω στα απλά δύο κτίρια. Μας απασχολούν το Square Meus, καταρχάς, στην πλατεία Meus, το οποίο χρειάζεται περισσότερο ε, ανακαίνιση και φυσικά εκένωση και δεύτερον ε, αποφασίσαμε ότι από τη νέα θητεία και μετά θα έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις για τους βουλευτές, αυτό έχουμε αποφασίσει κατά κανόνα, Χρειάζεται όμως και επιπλέον εμβαδών από το 2014 και την νέα θητεία, γιατί το κτίριο Τριμπέλ θα το έχουμε σε θέση μας μόνο από το 17 και μετά. Άρα πρέπει να βρούμε γραφεία για τους βουλευτές. Θα πάρουμε λοιπόν το κτίριο στην πλατεία Μέους υπαριθμών 8, Τα οικονομικά είναι καλύτερα εκεί από ό,τι είχε προταθεί προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον προηγούμενος ένικος. Έχουμε χαμηλότερο ποσοστό λοιπόν, χαμηλότερο κόστος για μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μετακομίσει το μεταξύ, έχει φύγει και έχουμε να κάνουμε με 25.000 τετραγωνικά μέτρα 38.000 πάνω από το 75 μάλλον τετραγωνικά χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος, ε, μάλλον συνολικά και τα 38.000 είναι πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και τα υπόλοιπα είναι κάτω. Στο υπόγειο δηλαδή. Θα έχουμε συνολικά στη σύμβαση για, από το 2014 και απέφυγα να σημειώσω στην ε, σύμβαση μίσθωσης τη δυνατότητα της τιμωρυθμικής αναπροσαρμογής. Έχουμε ένα μίστομα 7,6 εκατομμυρίων, δύο χρόνια δωρεάν, χωρίς δηλαδή μίστομα και συνολικά με συνυπολογισμό των δύο ε, αυτών ετών χωρίς ε, μίστομα, δωρεάν δηλαδή, το ποσό, το κόστος για μας θα είναι 7,6 εκατομμύρια, όπως σας είπα. Εδώ νομίζω ότι καλύπτουμε τις ανάγκες που είχαμε αναφέρει πριν από τρία χρόνια περίπου με ένα κόστος 300 ευρώ στο τετραγωνικό μέτρο. Είμαστε κάτω από τα 200 περίπου το τετραγωνικό και άρα είναι πολύ οικονομική πρόταση και ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα μισθώματα της περιοχής. Επιλέγουμε τη χρονομίστοση διότι μπορούμε έτσι να εξοικονομήσουμε από διάφορους φόρους και η συνολική τιμή είναι συμφέρουσα γιατί η αναπροσαρμογή των καλωδιώσεων, ανακαίνιση στο επίπεδο των καλωδιώσεων για τους υπολογιστές και τα λοιπά που θα μπορούσε να υπολογιστεί 8 με 10 χρόνια θα κρατήσει, θα αναπτυχθεί στα 12 χρόνια. Για δε αμίαντο και τα λοιπά δεν υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι γνωρίζω. Ευχαριστώ λέει η κυρία Χάουκαρα, δεν έχουμε γνώμη. Δεν, δεν, δεν, επιφυλάσσεστε ως προς το θέμα αυτό, καλώς. Όχι, άποψη έχω Πρόεδρε, απλώς επιφυλάσσομαι. Υπάρχει άλλο ένα Έγραφ, ε, κείμενο, κτίριο, αλλά πρέπει να το ξαναδιαπραγματευτούμε για να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε θα το αφήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια πρόεδρε της πολιτικής κτηρίων εν γέννη. Λοιπόν, εγώ έχω εξαντλήσει όλα τα θέματα τη ημερήσια διάταξη όσο με αφορά, αλλά πριν να αρχίσετε όλοι να τρέχετε έξω από την πόρτα. Τη Δευτέρα έχουμε Επιτροπή Προπολογισμών. Θα είδατε στο σχέδιο, στο σχέδιο ημερήσια διάταξη ότι υπάρχει περίπτωση να προβλεφθεί και συνεδρία συντονιστών. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται συνεδρία συντονιστών, αρκεί να την κάνουμε το το... στο Στρασβούργο. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή ε, ξεκούραση απόψε και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα στις 3.